Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Μπορούμε να ξαναρχίσουμε τη συνεδρία σας, παρακαλώ, με τις ανακοινώσεις του Προέδρου και την ε, ε, απόδοση των ε, πεπραγμένων από τις συνεδρίες των συντονιστών. Καταρχάς, οι συντονιστές συστήσαν την διαπραγματευτική εντολή για την έκθεση για την πρώτη αναθεώρηση της δέσμης των σιδηροδρόμων της κυρίας Σαρικιάνη. Η κυρία Σαρικιάνη λοιπόν <clears throat> μαζί με τους σκιώδεις εισηγητές έχουν εντολή για διερευνητικές συνομιλίες με θέμα όλες τις γνωμοδοτήσεις και μετά να ξεκινήσουν τον άτυπο τριμερή διάλογο επί τη βάση της πρώτης ανάγνωσης του Κοινοβουλίου με πλήρη υποστήριξη των σχεδόν εισηγητών και την υποχρέωση πλευράς της εισηγήτριας να επανέρχεται στους συντονιστές και να τους ενημερώνει τακτικά για τις εξελίξεις ως προς τους εισηγητές και συντάκτες νομοδοτήσεων. Οι αποφάσεις των συντονιστών έχουν τα εξή Ως εξής για την τροπολογία της, της ε, οδηγίας 126 2006 για τα άδειε οδηγήσεως για επαγγελματίες οδηγούς, όχι για τους ιδιώτες, με την ειδική αυτή κάρτα, ορίζεται ως ηγητής ο Πρόεδρος. Μάλλον από το Προεδρείο και επί τη βάση της εναλλαγής ε, των αντιπροέδρων στο Προεδρείο, ο, αποφασίστηκε το θέμα να αναλάβει η κυρία Τιτσάου γιατί είναι και πιο σχετικό με τον ταχογράφο που είχε προηγουμένω. Για το ε, θέμα των ελέγχων και πάλι έχουμε τις, ε, την εναλλασσόμενη ανάληψη από τις ομάδες, δηλαδή πάει στην ΚΟΕ. Μετά έχουμε το Περιφερειακό Ταμείο και την υποστήριξη για την εδαφική συνεργασία. Γνωμοδότης αυτή τη φορά και πάλι με σύστημα εναλλαγή, όπου σειρά έχει η Γκουε για άλλη μια φορά, άρα αναλαμβάνει και αυτή τη γνωμοδότηση. Διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές και ανάκληση της επαφάσεως 1364 πάει στο EFD, πάλι με το σύστημα της εναλλαγής. Υπενθυμίζω δε ότι αν μια ομάδα δεν θέλει να αναλάβει μια έκθεση τώρα σειρά τη, τη χάνει τη σειρά τη και πάει η τελευταία πάλι σειρά, αλλά η ΕΦΤ ανέλαβε να το, να το εκπονήσει. Η ανάκληση της αποφάσεως 1639 ανταγωνιστικότητα πλαίσιο, πρόγραμμα πλαίσιο, δημοσιονομική βοήθεια στο πλαίσιο των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ενεργείας αποφασίζεται να οριστεί από το ΕΛΚ ο εισηγητής. έγραφα προς ενημέρωση. Στα έγγραφα αυτά θεωρεί η ομάδα των συντονιστών ότι δεν χρειάζεται να τοποθετηθούμε ως προς την ετήσια έκθεση του 2010 για την εφαρμογή των κοινών κανόνων στην ασφάλεια των αέριων μεταφορών ή αντίστοιχα την ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θεσπίζει ένα σύστημα ε, διαχείρισης των αερομεταφορών Επίση, θεωρήθηκε ότι χρειάζεται να αντιδράσουμε στην ανακοίνωση προ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ένα πακέτο ανάπτυξη για, ε, για ολοκληρωμένε ευρωπαϊκέ υποδομέ. Διότι πρόκειται για ένα ζήτημα που ήδη καλύπτεται από το νομοθέτημα Connecting Europe. Όσον αφορά δε τη Single Sky, την νομοθεσία αυτή και την ε, νέα πρόταση θα συζητηθεί στους, στην προσεχή συνεδρία των συντονιστών και θα κριθεί ποια ομάδα θα είναι αυτή η οποία θα δώσει και το σχετικό πόντο. Πάντως αποφασίστηκε ότι θα είναι ε, έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας. Λοιπές νομοδοτήσεις, στόχοι του Κιώτο. Δεν αναλαμβάνεται δράση ανακοίνωση για την ε, ε, πρωτοβουλία για ευρωπαϊκά, για ευρωπαϊκά ομόλογα έργων, project, ε, Euro Project Bond. δεν αναλαμβάνουμε δεύτερη γνωμοδότηση, γιατί ήδη καλύπτεται από μία πρώτη που έχουμε αποφασίσει και έτσι δεν θα γίνει τίποτε περαιτέρω ανακοίνωση για το πλαίσιο μιας επόμενης γενεάς καινοτόμων χρηματοπιστωτικών μέσων ε, και πάλι δεν αναλαμβάνεται δράση. Μόνο τέσσερα έχουν μείνει ακόμα. Ανακοίνωση για τη στρατηγική διεύρυνση δεν αναλαμβάνουμε δράση ανακοίνωση για την υποψηφιότητα της Σερβίας. Δεν αναλαμβάνουμε δράση. Ανακοίνωση για μια σαφέστερη αντίδραση Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρόβλημα των ναρκωτικών. Δεν αναλαμβάνουμε δράση. Και ανακοίνωση, μάλλον έκθεση προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τα προβλήματα στις μεταφορές των ζώων Λένε οι συντονιστέ ότι είναι καλύτερο να περιμένουμε, να δούμε τι ε, επιλογές, ε, σε τι επιλογές θα προβεί η Γεωργική Επιτροπή και να αποφασίσει η Γεωργική Επιτροπή να συντάξει έκθεση, τότε και εμείς ως Επιτροπή Μεταφορών θα γνωμοδοτήσουμε. Το Connecting Europe εν τέλει ε, ενημερώνονται, ενημερώθηκαν οι συντονιστές για τις εξελίξεις προς την ε, πρόοδος εργασίας στο θέμα αυτό. Επιτροπολογία. Ο κύριος Ελκαντράου ενημέρωσε τους συντονιστές για τα ε, έγγραφα που δεν ε, παρουσιάζουν προβλήματα. Στην άλλη συνεδρία του Νοεμβρίου η άλλη συνεδρίαση μάλλον του Νοεμβρίου των ειδικών για το θέμα αυτό θα ετοιμάσει μια έκθεση που θα υποβληθεί στους συντονιστές το Δεκέμβριο, γιατί ξέρουμε ότι τους ενδιαφέρει. Στα διάφορα οι μέρες τέντη της Αμβέρσας. έχουν μια κορύφωση με τις ε, ομιλίες των συντονιστών που θα έχουν καθένα διαθεσία από 10 λεπτά. Και βέβαια θα κοιτάξουμε να συντονιστούμε ώστε όταν μιλάμε οι συντονιστές στην συνάντηση αυτή της Αμβέρσας να αποστέλουμε τα ίδια μηνύματα. Έχουμε επίσης από τον κύριο Μάλκον Χάρμπορ λάβει μια επιστολή για το θέμα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων πρόσκληση να συμμετάσχουμε στην εκδήλωση που θα η και εμείς θα ανταποκριθούμε με δύο γνωμοδοτήσεις για τα κύρια προβλήματα που εντοπίζονται στο θέμα αυτό. Το ένα είναι η, ε, τα δικαιώματα των ε, επιβατών και το άλλο είναι οι αδειοδοτήσεις και οι, άδειες, οι πινακίδες κυκλοφορίας ε, διαφορετικών κρατών σε, σε αυτοκίνητα, σε οχήματα που διασχίζουν τα σύνορα. Ένα άλλο πρόβλημα που μας απασχολεί επίσης είναι η πειρατεία, η θαλάσσια πειρατεία ιδιαίτερως, Έχει ετοιμάσει ο κύριος Βαντάλεν μια πρόταση και ζητούμε από τη γραμματεία να βοηθήσει ώστε να ε, γίνει μια περίληψη του κειμένου αυτού ώστε να μειωθεί στον απαιτούμενο βαθμό λέξεων σελίδων. Και είχαμε μια πρόσκληση από το Ευρωπαϊκό Εμπορικό Επιμελητήριο να επισκεφθούμε την ε, UPS στην Κολονία που συζητούν οι συντονιστές. Θα κοιτάξουμε να βρούμε μια ημερομηνία που να εξυπηρετεί όλους τους εμπλεκόμενους. Άρα συμφωνούν οι συντονιστές, απλώς πρέπει να βρούμε την κατάλληλη ημέρα για το είναι επίσκεψη αυτή. Επίσης, ε, ενημερωθήκαμε για μια επιστολή της Πολωνικής Προεδρίας για την πολιτική για το διάστημα τις πτυχές μεταφορών, δηλαδή που αφορούν την πολιτική την πολιτική. Και θεωρούν οι συντονιστέ ότι η συνεδρίαση τη 19η-21η Δεκεμβρίου δεν χρειάζεται να διαρκέσει τρει μέρε, θα περιοριστεί στις δύο πρωτες 19 και 20 Δεκεμβρίου δηλαδή. Αυτά είχα να σα πω από του συντονιστέ. Έχετε τίποτα άλλο εσείς να προσθέσετε, να συμπληρώσετε, να ρωτήσετε ή δάλλως. Φαντάζομαι ότι εγκρίνετε την ε, έκθεση των συντονιστών. Την έκθεση των εργασιών των συντονιστών καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Είναι οι στατιστικές καταγραφές ε, μεταφορών εμπορευμάτων οδικός. Νομίζω ότι δεν θέλετε να... δεν θέλει κανείς να ασχοληθεί με ένα τέτοιο θέμα, να περάσει ώρες βλέποντας τις στατιστικές ε, καταγραφές. Εν πάση περιπτώσει όμως είχαμε διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, επιτύχαμε συμφωνία ε, με το Συμβούλιο και την Κομισιόν ε, πάνω σε ένα συμβιβαστικό κείμενο το οποίο βρίσκεται στα, στους φακέλους σας. Όμως ε, θα σας πω ότι σε γενικές γραμμές συμφωνήσαμε ε, για την ε, προσαρμογή της παλιάς επιτροπολογίας σε κατεξουσιοδότηση πράξη. Βρέθηκε λοιπόν και μία συμφωνία όσον αφορά το εύρος καθώς επίσης και το περιεχόμενο της εντολής που, με την οποία θα η Επιτροπή. Ε, και βεβαίως εμείς θέλαμε πέραν αυτού να υπάρχει και η απαραίτητη ευελιξία αυτός ήταν και ο, ο στόχος της Επιτροπής Μεταφορών και ευρύτερα βεβαίως και του ιδίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βάσει και των τροπολογιών που υπέβαλε. Δεύτερον, όσον αφορά ε, τους ε, ε, ταχυγράφους και όσον αφορά ε, και τις ε, εκπομπές, βεβαίως εκεί είπαμε ότι θα πρέπει να προχωρήσει σε νέα αναδιατύπωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι το τέλος του 2014 ταυτοχρόνως δε θα πρέπει να αξιολογήσει ε, τα ευρήματα ε, όλων των ε, μελετών, κυρίως όσον αφορά των εκπομπών χερσαίων μεταφορών, λαμβάνοντας υπόψη διάφορες μεταβλητές. Τρίτον, δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων. Ήταν δικιά μας τροπολογία, τη δέχτηκε ε, το Συμβούλιο και δέχτηκε ότι η εξαίρεση θα γίνεται κάτ' εξαίρεση ε, σε ειδικέ περιπτώσεις και ε, λαμβάνοντας υπόψη ορισμένες γεωγραφικές ιδιαιτερότητες, ας πούμε, της Μάλτας. και μονάχα αργότερα θα αρχίσει να εφαρμόζεται ο κανονισμός στην Μάλτα οι ε, σκιώδεις συγητές στη συντριπτική τους πλειοψηφία στήριξαν τον ε, συμβιβασμό. Ε, δεχτήκαμε ότι το πνεύμα των τροπολογιών της Επιτροπής Μεταφορών ευρύτατα διαφαίνεται στο συμβιβασμό. Να ευχαριστήσω επομένως και τους σκιώδεις συγητές για την συνεργασία και να σας πω ότι θα υποβληθεί αυτός ο συμβιβασμός ως κείμενο τροπολογίας της Επιτροπής Μεταφορών στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου. Έχετε ερωτήσεις, η κυρία Λίχτεμπεργκερ παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για την πολλή δουλειά που κάνατε ε, για το θέμα αυτό. Είναι ένα σπάνιο παράδειγμα ε, της επιτυχίας που μπορούμε να έχουμε απέναντι στο Συμβούλιο και την ε, Κομισιόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδείξατε ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να αγωνιστεί και να πετύχει. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Όπως σας είπα, κάναμε πολλές συζητήσεις με τους σκιώδεις και οι σκιώδεις έπαιξαν πάρα πολύ με σπουδαίο ρόλο. Ε, κάναμε ωραία ομάδα. Είναι όλοι εντάξει, είναι όλοι ευτυχείς με την έκβαση των πραγμάτων. Πάρα πολύ ωραία. Επόμενο θέμα, ψηφοφορίες. Θα ζητήσω λοιπόν από όλους να πάρουν ε, τους, ε, τις καρτούλες τους, να είναι έτοιμοι Είστε όλοι έτοιμοι λοιπόν να κάνουμε ε, μία δοκιμή για να σιγουρευτούμε ότι δουλεύουν τα συστήματα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ναι, ναι, να ε, μετρήσουμε το ΕΛΚ. Εψήφισαν όλοι. will. Hang on, let's wait for Mrs. Mike. Ας περιμένουμε, γιατί η κυρία Μέσνερ φαίνεται ότι δεν έχει ακόμα ψηφίσει. Everybody Ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Είμαστε εντάξει. Στρέφουμε προς τη γραμματεία. Δεν πιστεύω να άκλεψε το ΕΛΚ να, να παραπανίσχοι. να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Γκρόση για τις προσπάθειες που καταβάλει έτσι ώστε να μην υπερβεί ο αριθμός των μελών του ΕΛΚ που ψηφίζει αυτή τη φορά. Έκθεση Σίμψον με μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνού Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορία τελική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Ομόφωνα. Επόμενο θέμα. Κατάλληλο ψηφοφορία για το χάρτη πορεία για έναν ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο μεταφορών, για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών. Έκθεση με ο Γκρό. Ε, θα ήθελα πριν ψηφίσουμε να σα πω ότι ε, υπήρξαν κάποια προβλήματα μετάφρασης και οποτεδήποτε ε, παρουσιάζονται τέτοια προβλήματα βεβαίως θα ελέγξουμε ε, την πιστότητα της μετάφρασης βασιζόμενη στο πρωτότυπο κείμενο. Ήθελα απλώς να καθησυχάσω όλους τους συναδέλφους ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Επίσης, υπομονή συνάδελφοι. γιατί εάν ε, καταπέσουν οι συμβιβασμοί θα έχουμε, τέλος πάντων, συμβιβασμός 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 40. Sorry? No, I, my says we vote on... Ε, σύμφωνα με το δικό μου κατάλογο ψηφοφορίας ψηφίζουμε για το 40. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβασμός 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 49. Τροπολογία debacker υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 44 υπέρ κατά αποχές μπορούμε να επαληθεύσουμε την τροπολογία 44 άρχεται η ψηφοφορία παρακαλώ ηλεκτρονική, ηλεκτρονικός έλεγχος εψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας <clears throat> και απορρίπτεται Συμβιβασμό 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμό 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμό 5. Συμβιβασμός 5. Ναι, καλά τα είπα εγώ. Συμβιβασμός 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 62 κανσιάν Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογ... Θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση. Εντάξει. Ελέγχουμε λοιπόν την τροπολογία 63. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. Τροπολογία 66 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 65 έχει αποσυρθεί, επομένως συμβιβασμός 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 71. Ε, τροπολογία Βαντάλεν. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 72. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 74 τέσσερα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 78 όχι, καταπίπτει. Ε, μονάχα η διαγραφή ε, της τροπολογίας 78 καταπίπτει, επομένως ψηφίζουμε το υπόλοιπο. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Το ίδιο νομίζω και με την τροπολογία 80, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ε, συμβιβασμός 8, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβασμός 9. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 115 της κυρίας Αγιάλα Σέντερ. Παρακαλώ κυρία Αγιάλα Σέντερ. <clears throat> Μισό λεπτό να βάλω και τα ακουστικά μου. Α, να ζητήσω μια ερώτηση. Μια ερώτηση. Ε, λοιπόν, είναι ένα σημείο το οποίο αφορά μόνο τα λογιστικά στοιχεία. Ουσιαστικά να παραμείνει αυτό το φόρουμ ε, logistics. Νομίζω ότι συμφωνείτε να μην καλυφθεί αυτό το θέμα από τις συμβαστικές προτάσεις, αλλά βλέπω ότι δεν υπάρχει συμφωνία αυτή τη στιγμή. Απλά Σα υπενθυμίζω ότι είχε γίνει ένα σχόλιο χθε ότι θα το στηρίζατε. Αυτό το φόρουμ λοιπόν συζήτηση ε, και προτάσεων για την εφοδιαστική, για το logistics, ε, θέλουμε να παραμείνει. Αυτό θέλω να σα υπενθυμίσω. Εντάξει, δεν θα κάνουμε τώρα ολόκληρη συζήτηση, ε, αλλά εν πάση περιπτώσει ψηφίσουμε την 115 για άλλα σέντερ υπέρ. Κατά αποχές ε, ηλεκτρονική επαλήθευση επί της 115. Κύριε Γκρός, πριν από το ηλεκτρονικό έλεγχο. Κύριε Γκρός. Θα πρότεινα, Πρόεδρε, να μείνουμε βέβαια στον κατάλογο των ψηφοφοριών, να τον ακολουθήσουμε, αλλά με τα όσα είπε η κυρία Γιάννα Σέντερ, να, προσαρμοστούμε σε μια ε, διατύπωση που θα πάει στην Ολομέλεια, έτσι ώστε να υπάρχει Okay, Ας ψηφίσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 115 Αγιάλα Σέντερ. Ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Και εγκρίνεται έτσι κι αλλιώς. Θα το αναφέρετε στην ε, Ολομέλεια. Τροπολογία 117. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο, μετά από το Energy Supply μέχρι το τέλος, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 119 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 123 υπέρ, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση, ωραία, επί της 123, παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Και απορρίπτεται. Συμβιβασμός 10. Χωρίς μικρόφωνο, δυστυχώς δεν ακούμε. Όχι. Ε, για μένα ήταν ε, σαφές ε, και το εδήλωσα. Επομένως τελειώνει η συζήτηση. Συμβιβασμός 10. Γιατί διαφορετικά θα αρχίσουμε να ξανασυζητάμε όλες τις τροπολογίες. Λοιπόν, ψηφοφορία κατά τμήματα. Πρώτον μέχρι το added value υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα είναι το υπόλοιπο της τροπολογίας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 11. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 131. Ερτογ υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 133 τικάου υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 139 Bradburn υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 141 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 140 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 142 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 143 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 144 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ωραία. Τροπολογία 144. Ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται. Ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβιβασμός 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 150 υπέρ κατά αποχές θα το ελέγξουμε γιατί δεν είδα καλά το αποτέλεσμα. Άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία από τις τροπολογίες 150. Νομίζω πως απορρίπτεται, αλλά δεν είμαι και σίγουρος. Η πολιτική μου ομάδα δεν σήκωσε καλά τα χέρια της. Λοιπόν, πέρα της ψηφοφορίας και απορρίπτεται. 151 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 152 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 153 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 156 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση της 156 ψήφισαν όλοι Πέρας της ψηφοφορίας. Και εγκρίνεται. 160 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 176. 176 και συγκατανεύει και ο Ματιό, οπότε όλα καλά. Απορρίπτεται η 176. 177 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, συνδυασμός 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 186 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 188 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβασμός 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβιβασμός 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 217 τρεμόζο ή μπαλτσέλς υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2.32. 2.32, κράμερ και λοιπόν, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.34, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2.35, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβασμός 20, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 2.44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2.49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, συμβιβασμός 23 υπέρ κατά αποχές θα ήθελα να ελέγξουμε ε, συμβιβασμό συγγνώμη 23 άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρασε και εγκρίνεται. Τροπολογία 258. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 259. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 260. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 261. 260, ε, α, για το 260, ωραία, άρχεται η ψηφοφορία. ε, ψήφισαν όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Και απορρίπτεται. 261 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, ε, ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφοφορία λοιπόν ηλεκτρονική για την 261 άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρασε. και εγκρίνεται. Συμβιβασμός 24 σε τέσσερα τμήματα από ό,τι βλέπω. Ένα, δύο, τρία και... Ε, ε ας ξεκινήσουμε πρώτα με την ορτορική σκέψη Ένα, Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δύο, Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τέσσερα, Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Το υπόλοιπο του κειμένου υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δύο εξήντα τέσσερα Bradburn υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 269 το πρώτο τμήμα της τροπολογίας μέχρι εκεί που λέει safety objectives. Ψηφίζουμε λοιπόν γι' αυτό έχει αποσυρθεί και επομένως ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα της αρχικής τροπολογίας 269 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 271 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 272 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 273 και 274 έχουν καταπέσει. 284 λοιπόν ψηφίζουμε υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 286 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 286 υπέρ. Κατά θα ελέγξουμε. Θα ελέγξουμε λοιπόν 288. Ε, 288 άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρα της ψηφοφορίες. Απορρίφτεται. 289 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός 25 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 300. Χωριστή ψηφοφορία, κατά τμήματα λοιπόν. Το πρώτο τμήματα μέχρι ε, Transport and Logistics Operation. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της τροπολογίας, υπέρ, κατά, αποχές. Μπορούμε να ε, κάνουμε μια ηλεκτρονική επαλήθευση για την ψηφοφορία του δεύτερου τμήματος. Ψήφισαν όλοι πέρα της πληροφορία. Και εγκρίνεται επομένω και το δεύτερο τμήμα. Τροπολογία 303 της κυρίας Μπιλμπάου υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 306 Wills υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβασμός 26α υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 26β. 26β λοιπόν υπέρ. Ηλεκτρονική επαλήθευση. 26β συμβιβασμός. Εψήφισαν όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. Και απορρίπτεται. Άρα τι κάνουμε τώρα, λέει ο πρόεδρος. Τρία σαράντα έξι. Τρία σαράντα έξι. This is the port services bit. My advice is Εάν δεν έχει εγκριθεί ο συμβασμός 26β, θα πρέπει να ψηφίσουμε την 306, 307, 8 και 9 που, είναι, που αφορούν ακριβώς την διαγραφή αυτής, της, ε, αυτού του τμήματος. 306 λοιπόν. Η... Θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τις πιο μακρινές τροπολογίες. Άρα θα πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτές που ζητούν διαγραφή. Πού είναι η 346 όμως, στον ε, κατάλογό μου εδώ. Got it. Right. 346 Φλέκενστάιν. Υπέρ κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση. Νομίζω πως εγκρίνεται, αλλά επειδή είναι σημαντική τροπολογία να είμαστε σίγουροι. 3.46 ψήφισαν όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας και εγκρίνεται. 309. 309. Ουτζίας ε, για την παράγραφο 16, Παύλα 1, 309. Ουτζίας υπέρ κατά Αποχέσε. απορρίπτεται. 305. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3.20 Έρτογκ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3.22 της κυρίας Μπιλμπάου υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. <laughs> Uh, just a question, sir. Μια ερώτηση. Τροπολογία 351 Higgins. Δεν την ψηφίσαμε αυτή την τροπολογία. Όχι. Μια και απερίφθη ο συμβιβασμός 26β, ε, ξεκινήσαμε από την τροπολογία 309, η οποία, ε, η οποία ε, κάνει, προχωράει σε διαγραφή και μετά πηγαίνουμε από τις πιο απομακρυσμένες στις πιο κοντινές. Ναι, ναι, δεν το κατάλαβα αυτό. Ωραία. Η τελευταία λοιπόν που ψηφίσαμε απερίφθη, 322, 309, προφορική τροπολογία και το κείμενο αναφέρεται σε χωριστή στήλη. Ψηφίζουμε λοιπόν μαζί με την προφορική τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 342, again with ε, Επόμενη τροπολογία με την προφορική τροπολογία Καντσιάνα. Ε, υπάρχει, ε, αναφέρεται στα eco bonus, στα οικολογικά bonus υπέρ κατά νομίζω ότι θα πρέπει να ελέγξουμε 3.42 με την προφορική τροπολογία. Τροπολογία Καντσιάν. Ε, πέρας της ψηφοφορίας. Και απορρίπτεται. Γιατί είναι 20 υπέρ, 20 κατά. Απορρίπτεται λοιπόν. 345 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Την 346 την έχουμε ήδη ψηφίσει, ήταν η πρώτη. Άρα συμβιβασμός 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 373 Κράμερ, Λίχτεμπεργκερ και λοιπόν υπέρ, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 381 έχει ήδη καταπέσει γιατί ο συμβασμός 15 εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 28 υπέρ. Α, ναι. Υπάρχει και μία προφορική τροπολογία που έχουν ζητήσει οι πράσινοι στην Παύλα 4. Έχετε όλη την προφορική τροπολογία. Πολύ ωραία την αμφισβητεί κανεί όχι. επομένω συμβιβασμό 28 με την προσθήκη τη προφορική τροπολογία υπέρ. Ε, να κάνουμε, ε, μάλλον να ξεκινήσουμε από την αρχή. Συμβιβασμός 28 με την προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πώς είπατε? No, we voted it with the oral amendment, yeah. So, we now go to 386. 386. Υπέρ. 386. 386. Τροπολογία 386. Παράγραφος 18, Παύλα 1α νέο. Και η πράσινη είναι έτοιμη. Ναι, κατανοώ ότι υπάρχει μια δυσκολία γιατί είναι μπερδεμένα όλα αυτά τα πράγματα. Τροπολογία 386 της κυρίας Μπιλμπάου υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 398 ε, με την και η 402 γιατί είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 40 υπέρ. 400 συγγνώμη υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 401 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 403 υπέρ. 403 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 407 υπέρ. Κατά αποχές. Ε, θα ήθελα να κάνουμε και μια ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία αυτή. Άρχεται η ψηφοφορία επί της 407 ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Και απορρίπτεται. 412 της κυρίας Τικάου υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση 412 δεν ήταν σαφές το αποτέλεσμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Και εγκρίνεται. 413 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 επί της σκέψης 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 ε, ψηφοφορία κατά τμήματα. Το πρώτο τμήμα θα είναι μέχρι εκεί που λέει for decision making within this field και το δεύτερο τμήμα βέβαια θα είναι το υπόλοιπο. ε, ψηφοφορία επί του πρώτου τμήματος υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβασμός 30 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 7 για την αιτιολογική σκέψη Β του κυρίου Τρεμόζα Ιμπαλσέλς. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 της κυρία Μπιλμπάου. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 18, ψηφοφορία κατά τμήματα, δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα EU Regions, δεύτερο τμήμα το υπόλοιπο. Η πρώτο τμήμα της 18 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται επίσης. Τροπολογία 19 του κ. Κόχ υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ κατά αποχές εν, απορρίπτεται. Τροπολογία 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. «29 απεσύρθη, 30 καταπίπτει, τροπολογίες της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Ευτυχώς πολλές έχουν καταπέσει ήδη. Δεν το είπα αυτό και κανείς δεν το άκουσε. Έτσι κι αλλιώς ε, με θεωρούν πολύ κακό παιδί, μη μάθουν και τίποτα τέτοιο. Τροπολογία περιβάλλοντος 3, NV3. Ε, επί της παραγράφου 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. NV4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Φτάνουμε τώρα στην NV7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. NV8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Νομίζω ότι επόμενα πρέπει να ψηφίσουμε για την παράγραφο 26. Η 22 καταπίπτει λόγω του ότι η 160 έγινε δεκτή. Παράγραφος 26, NV26. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 28, 28 ένβη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ένβη 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Πάμε τώρα στις τροπολογίες της Επιτροπής Ήτρε. Ήτρε 2. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται ή 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήτρα, ήτρε 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, τροπολογίες της Reggie, Reggie 2 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, Reggie 7, Reggie 4 μάλλον, Reggie ναι, 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, τώρα ψηφίζουμε τη Reggie 7, Α, όχι, πρέπει να ψηφίσουμε και τη Ρέτζι 6, γιατί η 261 δεν ψηφίστηκε. Υπέρ, κατά, αποχές. Ε, θα ήθελα να ελέγξουμε λίγο την ψηφοφορία για την ε, τροπολογία 6 της Επιτροπής ε, Ρέτζι. Ψήφισαν όλοι, πέρασε. Και απερίφθη. Ρέτζι 7, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εψήφισαν 41, 34 ψήφοι υπέρ, 5 ψήφοι κατά, 2 αποχές. Συγχαρητήρια κύριε Γκρός. Right, next. Λοιπόν, Επόμενο λοιπόν θέμα. Ναι. Right, we now go on to the PNR. Γνωμοδότηση Λίχτενμπεργκερ για τα δεδομένα PNR. Δύο τροπολογίες έχουν αποσυρθεί. 65 και 163. 65 και 163 λοιπόν πάνε. Αν είναι στο καταλογό σας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την ε, τροπολογία 7 και αντίστοιχα σημεία 8 και 2 υπέρ, αμπλόκολες αυτές, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Επόμενη ομάδα, το κομμάτι Terrorist Offenses and Serious Transnational Crime. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Εντάξει, να το ελέγξουμε, άρχεται η ψηφοφορία. Ματιέ, μόνος έμεινες νομίζω. Αν ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας, εδώ και το αποτέλεσμα. 26 υπέρ 15 κατά εγκρίνεται. Επόμενη ψηφοφορία επί της τροπολογίας 7 και 61 που είναι ταυτόσιμες ψήφι υπέρ κατά αποχές να το ελέγξουμε. Τροπολογίες 7, 61. 7 και 61. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Εγκρινώνται. Τροπολογία 62 Bradburn Ψήφι Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται, αλλά θέλετε να το ελέγξουμε, ας το ελέγξουμε. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται πράγματι. συγκρατήσω, Φίλιπ. Λοιπόν, επόμενη. ...63 και 64 τροπολογίες με την προφορική τροπολογία. Συμφωνείτε όλοι ωραία. Λοιπόν, ψήφι Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε Τη τροπολογία 63 63-64 συν προφορική τροπολογία άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Και αυτές συγκρίνονται. Επόμενη. Τροπολογία 67, τροπολογία 68, τροπολογία 69. Ταυτόσιμες. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Άρα πηγαίνουμε στην τροπολογία 71. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2F. Συμφωνή. Push method. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άρα οθούμε, πιέζουμε και δεν έλκουμε. Λοιπόν, τροπολογία 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 15 αρχή αναλογικότητας principle of proportionality υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβιβαστική για το άρθρο 2 παράγραφος 1 Serious Transnational Crime. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 87 τικάω υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογίες 88 και 89 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 9 που εισηγητή υπέρ, τη εισηγητρίας υπέρ, κατά αποχές να ελέγξουμε την τροπολογία 9 παρότι θα έλεγα ότι απορρίπτεται. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Ένας παραπάνω για το ΕΛΚ. Ματιέ. Λοιπόν, ψηφίσατε όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογίες 90 και 91. Πρέπει να τις ψηφίσουμε τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Τροπολογία 92. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 93 μαζί με την 94. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία τώρα 96 και 97 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται και αυτές. Ας ελέγξουμε, εντάξει. 96 και 97 έρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρα ψηφοφορίας. 22 υπέρ, 20 κατά εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4. Danger in delay. Άρχεται. Όχι. Λοιπόν, υπέρ. Κατά. Εποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Αλλά εκ νέου θα προτιμήσω να το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για τη συμβιβαστική 4. Danger in delay. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται συμβαστική 4. Εκατό και 101 τροπολογίες. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε. Αν και θεωρώ ότι απορρίπτονται. Ελέγχουμε τις 100-101. Άρχεται η ψηφοφορία. Η 98 έχει καταπέσει πάλι πιο πολλές ψήφοι από ό,τι πρέπει για το ΕΛΚ. Λοιπόν, πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται, εγκρίνονται. Συμβιβαστική 6. Χωριστή ψηφοφορία για την παράγραφο 3 έχει ζητήσει η ομάδα των συντηρητικών. Πρώτα λοιπόν παράγραφος 3 της συμβαστικής 6. Επέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το υπόλοιπο τώρα της συμβαστικής υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και επομένως πηγαίνουμε τώρα στην τροπολογία 114 και στην τροπολογία 117. Ψήφι υπέρ, κατά. Ελέγχουμε τις τροπολογίες 114 και 117 άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρας. Απορρίπτονται. Περνάμε λοιπόν τώρα στην τροπολογία 115. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 116 είναι γλωσσικής υφής. Δεν την ψηφίζουμε. Πηγαίνουμε στην τροπολογία 11 τις εισηγήτριας γιατί οι υπόλοιπες καταπίπτουν. Ψήφι υπέρ τις 11. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 138 πύρκερ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12 της εισηγήτριας υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογίες 143 και 144 ταυτόσιμες τροπολογίες ψήφι υπέρ. Κατά αποχές να ελέγξουμε τις δύο αυτές τροπολογίες 143-144. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε ψηφοφορίας. εγκρίνονται. Τροπολογία 13 και 14. Μπλοκ. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Πηγαίνουμε από ό,τι νομίζω τροπολογία 150. Έτσι, σωστά, ωραία. Μαρ Σινκίεβιτς, ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 151. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 15 της εισηγήτριας. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία χωρίς το τρίτο τμήμα, γιατί έχει καταπέσει. Τροπολογία 153 άνευ του τρίτου τμηματο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ελέγχουμε. Ελέγχουμε. Τροπολογία 153 τικά χωρίς το τρίτο τμήμα άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 152-154. Το τελευταίο του τμήμα που είναι ταυτόσιμο είναι το μόνο που θα θέσω σε ψηφοφορία. At the latest at the end. Ως προσθήκη στην τροπολογία 15. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 159 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 155 χωρίς το τελευταίο τμήμα που έχει καταπέσει. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 157 χωρίς το τελευταίο τμήμα. Α, όχι, έχει καταπέσει. Επειδή εγκρίθηκε 155, άρα πηγαίνουμε στην 158 Μαρκιντσίβης. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 120, 160, συγγνώμη, υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 16 της εισηγητρίας, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογίες 162-164, ταυτόσιμες τροπολογίες υπέρ, κατά, απο, εγκρίνονται. 166-167 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται. 168-169 ψήφι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 170. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Έως εκεί που λέει PNR data. Ψήφι υπέρ. κατά, αποχές, να ελέγξουμε το πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία, πρώτο τμήμα της 170. Ψηφίσατε όλοι, πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα τώρα, δεν ξέρω αν έχει νόημα να ψηφίσουμε το υπόλοιπο του κειμένου. Έχει, λοιπόν, θέτω σε ψηφοφορία δεύτερο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 171 Σμιτ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 172. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 17 της γήτριας. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογίες 173, 174, 176. Ναι, μεν ταυτόσιμες, αλλά έχουμε ψηφοφορία κατά τμήματα. Το πρώτο τμήμα είναι διαγραφή του κομματιού από το upon the date ως article 6.1 are collected. Υπέρ, κατά, αποχές να ελέγξουμε. Πρώτο τμήμα των 173, 174, 176. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα. Της 173 διαγραφή του κομματιού από Until Two Years μέχρι άρθρο 6.1. Are collected. Article 6.1. Ε, are collected. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. άποχες θα ελέγξουν. Δεν ξέρω τι έκανε το ΕΛΚΑ, τι ψήφισε. Άρχεται η ψηφοφορία, δεύτερο τμήμα. Ψηφίσατε όλοι πέρας. Εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα. Τρίτο τμήμα. Διαγραφή του κομματιού Member States έως πάλι are collected. Υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Άρα, 175 καταπίπτει. Εγκρίναμε το δεύτερο τμήμα της 173, άρα καταπίπτει 175 και πηγαίνουμε στην 177. Λοιπόν, 177 και 178 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 18 της υπέρ, κατά, αποχές ελέγχουμε τη 18. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται με ισοπαλία, ισοψηφία. 180 και 181 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 182 και 183 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε. Τις 182, 183 έρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτονται. Τροπολογίες 184-185 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 186-187 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 188-189 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 190-191 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 192-193 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 194-195 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 196 τώρα δεν ξέρω, έχει καταπέσει, όχι, 196 Bradburn υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 197 μαζί με την 198 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται 199 200 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται 201-202 τροπολογίες υπέρ. Κατά αποχές. Ας ελέγξουμε τις δεύτερες τροπολογίες 201 και 202. Αν ψηφίσατε όλοι, Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτονται. Συμβιβαστική για το σημείο 12 του παραρτήματος. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογίες 206 και 207 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε παρακαλώ τις 206 και 207 έρχεται η ψηφοφορία. Αν ψηφίσατε όλοι, πέρασε. Απορρίπτονται 208-209 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται τροπολογίες 2-10-2-11 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται 2-12-2-13 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται. 2.14-2.15 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. Να ελέγξουμε. Καλώς. 214-215 έλεγχος. Ψήφισατε όλοι. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίφθηκαν. Προπολογίες 216-217. Υπέρ. Κατά αποχές ελέγχουμε και αυτές τις δύο τροπολογίες 2.17-2.18 άκτη ψηφοφορία. 2.16-17 συγγνώμη, πέρας ψηφοφορίας απορρίπτονται τροπολογίες 2.18-2.19 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε, ελέγχουμε μάλλον το ίδιο αποτέλεσμα θα έχουμε άρχεται η ψηφοφορία πάντως ψηφίσατε όλοι πέρας Πράγματι ήταν το ίδιο αποτέλεσμα. Απορρίπτονται με ισοψηφία. Τροπολογία 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε την τροπολογία 19. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Πράγματι με στρεπτική πλειοψηφία 36 ψήφι υπέρ 5 κατά. Ξέρω ότι είναι πολλές ψηφοφορίες, αλλά βοηθήστε μας λιγάκι σηκώνοντας χέρια παρακαλώ. Πού πηγαίνουμε τώρα. Στην 20 τροπολογία. ΣΜΙΤΑ, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται τροπολογία 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε την τροπολογία 1 που νομίζω ότι εγκρίνεται. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Πράγματι εγκρίνεται. Συμβιβαστική R11. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 26, 27, συγγνώμη και 28. 27 και 28 υπέρ. Κατά εποχές ελέγχουμε τις 27-28. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίφθηκαν. Τροπολογία 29 ρικέ. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογίες 31-32 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε την 34 παρακαλώ. Τροπολογία Σμιτ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 35. De Grandes. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 36 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 37 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική R15 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 42 κοντεύουμε Κοντεύουμε. Τροπολογία 42. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 43. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 44. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 45. Υπέρ κατά αποχές. Να ελέγξουμε παρακαλώ την τροπολογία του κυρίου Σμίτ παριθμό 45. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την 46 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 47, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ας περάσουμε στις 5, 48, 49 και 50. 5, 49, 50. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Τροπολογία 52. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 53. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, απορρίπτεται. Τροπολογίες 55 και 57 είναι ταυτόσιμες. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε παρακαλώ τις τροπολογίες 55 και 57. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. εγκρίνονται. Τροπολογία 54. Ψήφι Κατά αποχές απορριπτώνται. Τροπολογία 56 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 25 ψήφοι υπέρ 15 κατά μια αποχή εγκρίνει η γνωμοδότηση της κυρίας Λιχτεμπέργκερ την οποία και συγχαίρουμε. Πάρα πολύ καλά τα καταφέρατε σε ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα. Και τώρα έχουμε την έξι κυρίας Wills για την φορολόγηση προϊόντων, ενεργειακών προϊόντων και ε, ηλεκτρικής ενέργειας. Ξεκινώ με την τροπολογία υπαριθμών 11 του κυρίου Κοχ. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ας επαληθεύσουμε την 27 της κυρίας Τετσάου, παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε φορές. Έλα, Μάικλ. Εντάξει, ο κύριος Κράμερ λοιπόν θέλει να καταψηφίσει. Προχωρώ στην 28, ο κύριος Ρικέ υπέρ του κύριου Ρικέ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 30. Καταπίπτει. 29 καταπίπτει. 31 καταπίπτει και πάμε στην 5 ε, τώρα του εισηγητού υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. Κύριε Γουίλς. Θα ήθελα, Πρόεδρε, για την υπαριθμόν 5 τροπολογία να πω ότι 6, 7 και 8 μπορούν να αποσυρθούν. Και επίση αποσύρεται και η διαγραφή στο 4 και στο 10. Ευχαριστώ κύριε φίλη. Αποσύρεται λοιπόν την 6, την 7, την 8 και επίσης αποσύρεται τις ε, προτάσεις διαγραφής στις τροπολογίες 4 και 10. Τελευταία, τελευταία. Καλώς. Ευχαριστώ και περνούμε στην 34 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 35 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 36 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 37-38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 10 με την ε, απόσυρση της διαγραφής υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 41 Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 12. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά επαληθεύουμε παρακαλώ και 14 εψήφισαν όλοι εντάξει απορρίπτεται 15 υπέρ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 όχι, έχει καταπέσει το δεύτερο και ψηφίσουμε το πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 26. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 24. Με τεχνική προσαρμογή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 25 υπέρ, ε, καταπίπτει μάλλον, καταπίπτει 25 και πάμε στην 4 χωρίς την διαγραφή. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται με 31 ψήφους υπέρ, 9 ε, ναι, ψήφους κατά και μία μόνο αποχή. Συγχαρητήρια κυρία Μίλης. Αγαπητοί συνάδελφοι, έτσι ολοκληρώνονται οι ψηφοφορίες μας. We have a little bit. you? It's a little bit early. Are you ready? Κυρία Σάβισαρ, ξέρω ότι έχουμε ότι είμαστε λίγο πιο νωρίς από ό,τι είχαμε προβλέψει, αλλά αν είστε έτοιμοι να κάνουμε την παρουσίαση. Προτείνω, αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ, να ακούσουμε την έκθεση κυρία Σάβισαρς και έτσι μετά να δούμε και την παρουσίαση της εκθέσεως για την βιώσιμη κινητικότητα που θα χρειαστεί να ξεκινήσει μόνο στις 11.30 όπως έχουμε προβλέψει. Άρα ας δούμε την κυρία Σάβησα πρώτα. Και αν μπορέσουν οι κλητήρες μας να δούμε τι έγινε αυτό το τσάι το χάσαμε το τσάι μας. Τι έγινε. Όποιος αποχωρεί, παρακαλώ, ας αποχωρήσει τώρα. Ήσυχα. Μετάξει. Ναι, εντάξει. Επόμενο θέμα λοιπόν στην ημερήσια διάταξη. Έχουμε την περιεκτικότητα των καυσίμων πλοίων σε θείο σχέδιο γνωμοδότησης της κυρίας Σάβησαρ, η οποία έχει και το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρόκειται για ένα σχέδιο γνωμοδότησης προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, το οποίο σχετίζεται με την τροποποίηση της οδηγίας για το περιεχόμενο καυσίμων πλοίου πλοίων σε θείο και θα έχει σημαντικέ ε, συνέπειε προ την πολιτική των μεταφορών. Θα ήθελα ξεκινώντα να σα πενθυμίσω ότι ανεξαρτήτω ε, τη έκβαση τη δική μα δουλειά και τη ε, δουλειά τη Επιτροπή του Περιβάλλοντο, έχει καταλήξει σε συμφωνία η διεθνή Ναυτιλιακή Οργάνωση το 2008 και τίθεται αυτή η συμφωνία ενισχύ. Πρόκειται δηλαδή για μια συμφωνία η οποία ορίζει νέες οριακές τιμές ε, για την περιεκτικότητα των καυσίμων πλοίων στις θείου, στις περιοχές ελέγχου των εκπομπών θείου. Με άλλο το όριο από 1,5% 1% από 1η Ιουλίου 2010 και 0,1% από 1η Ιανουαρίου 2015. για τις περιοχές ελέγχου των εκπομπών θείου. ΠΕΘ. Πέραν αυτών των περιοχών ελέγχου των εκπομπών, τα όρια είναι από 4,5% σε 3,5% από 1η Ιανουαρίου του 2012 και 0,5% από 1η Ιανουαρίου του 2020. Εμείς όμως ως προ την συγκεκριμένη αυτή προδιαγραφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουμε συγκεκριμένη ε, διάταξη. Θα μπορούσαμε να καθυστερήσουμε την εφαρμογή των νέων προδιαγραφών ε, του 2020, δεδομένου ότι ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός ε, ΔΝΙ σκοπεύει να προβεί σε μια αναθεώρηση και άρα ίσως χρειαστεί μετά το 2015 να ισχύσουν νέες οριακές τιμές στις συγκεκριμένες περιοχές. Εάν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προβεί στις σχετικές ε, ε, προσαρμογές, δεν θα έχουμε τους κανόνες που ε, θα ευθυγραμμίζονται με τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου. Θα έχουμε διαφορετικά μέτρα και σταθμά. Έτσι λοιπόν, Εάν δεν περιοριστούν οι οριακές ε, τιμές για το θείο, θα έχουμε υψηλότερη αναλογία θείου στις θαλάσσιες μεταφορές από ό,τι στι χερσαίες. Και η, διαφορά, η απόκληση μπορεί να αγγίξει και το 72%. Δεύτερον, Ε, η μείωση αυτών των ε, εκπομπών ασφαλώς θα βελτιώσει και ε, θα βοηθήσει σημαντικά στη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθήκων. Ξέρουμε ότι οι εκπομπές θείου είναι υπεύθυνε για πολλούς πρόωρους θάνατου, για χιλιάδες πρόωρων θανάτων στην Ευρώπη καθέτος. Επίσης, η εισαγωγή αντίστοιχων ορίων ανά τον κόσμο θα βοηθήσει βέβαια στην εξασφάλιση ενός ισότιμου πεδίου ανταγωνισμού σε ολόκληρο τον κόσμο. Για τη συγκεκριμένη λοιπόν πρόταση που έχω διατυπώσει στη γνωμοδότησή μου. Έχω ζητήσει από όλες τις πολιτικές ομάδες ε, να καταθέσουν τις ε, τοποθετήσεις τους, τις προτάσεις τους. Δυστυχώς όμως δεν κατέστη δυνατό να συγκεράσω τις θέσεις αυτές σε μία που να ικανοποιεί όλες τις, ε, άλλες, όλες τις πολιτικές ομάδες στο ίδιο, στον ίδιο βαθμό. Έτσι λοιπόν αναγκάζομαι να ακολουθήσω την επιλογή των ΗΠΑ και του Καναδά που ορίζουν ως όριο απόστασης τα 2.000 ναυτικά μίλια και αυτό έχω περιλάβει στην ομοδοτήσή μου. Ξέρω ότι υπάρχουν αμφιβολίες για το κατά πόσον θα έχουμε των 200 ναυτικών μιλίων κατά πάσα πιθανότητα. Ε, ξέρω ότι έχουμε βέβαια αμφιβολίες για το κατά πόσον θα είμαστε έτοιμοι το 2015 για την προσαρμογή αυτή ως προς τα κάψιμα που θα χρησιμοποιούν τα πλοία. Ξέρω ότι θα είναι δύσκολο, αλλά από την άλλη έχει έρθει η ώρα να ε, πάρουμε αποφάσεις. Και από την απόφαση του Διεθνούς Αυτιλιακού Οργανισμού του 2008 δεν έχει προχωρήσει τίποτα άλλο, δεν έχει παρισφρήσει κάποια άλλη ε, εξέλιξη και υπάρχουν κάποιοι που γνωρίζουμε ότι θέλουν να παγώσουν οποιαδήποτε εξέλιξη. Ωστόσο, Πιστεύω ότι μετά το 2018 καλό θα είναι να μην βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση οι επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες έκαναν προσπάθεια για προσαρμογή στην ε, νομοθεσία ε, και που όμως τελικά δεν μπορούν να, να τηρήσουν αυτές τις διατάξεις μόνο και μόνο γιατί δεν υπάρχουν ε, διαθέσιμα καύσιμα της ποιότητας που ορίζεται. Υπάρχει η δυνατότητα να ε, αναμειχθεί το πετρέλαιο με υγροποιημένο φυσικό αέριο, LNG. Αυτό θα επιτρέψει στι αμφιλιακέ εταιρείε να επιλέγουν τον οικονομικότερο τρόπο συμμόρφωση προ οριακέ τιμέ, λαμβάνοντα υπόψη την ηλικία και των σκαφών, καθώ και τι διαδρομέ για το. Ε, τις διαδρομές που αυτά αναμένεται να εξυπηρετήσουν. Πάντως πιστεύω ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεδομένου ότι και αυτά θα επωφεληθούν από την τήρηση των διατάξεων. Τα ωφέλη για τη δημόσια υγεία θα είναι πολύ υψηλότερα από το προβλεπόμενο κόστος. Άρα πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει η προσαρμογή τα μέτρα αυτά δηλαδή θα είναι αποφελή προς τους πάντες, προς το, για το περιβάλλον μας, για την εξασφάλιση ενός ισότιμου πεδίου ανταγωνιστικής αναμέτρησης και με όρια 2% για τα εμπορικά πλοία και 1,5% για τα επιβατηγά, πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε ικανοποιητικές ε, διατάξεις. Αυτό με δεδομένο ότι ε, δεν θέλουμε να, προ, να προξενήσουμε μετακύληση των φορτίων αυτών από τις θαλάσσιες οδούς στις χερσαίες οδούς, γιατί αυτό βέβαια θα αντέβαινε στον σκοπό των ίδιων της οδικής. Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σας. Ευχαριστώ πολύ αγαπητή συνάδελφοι. Ο κύριος Κούν, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Σάβησαρ για, το, για την έκθεση αυτή, για την ομοδότηση αυτή που επεξεργάστηκε με τόσο πολύ ε, προσοχή στον χώρο των βορείων ακτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2015 Ε, ξέρουμε ότι θα υπαχθούν στις λεγόμενες ΠΕΦ, δηλαδή περιοχές ελέγχου των εκπομπών θείου. Πρόκειται για τη Βόρεια Θάλασσα, για τη Βαλτική, για, την Ανατολική, τις ανατολικές ακτές των Βρετανικών νήσων και τη μάχη σε ένα βαθμό. Και έτσι πολύ σωστά η κυρία Σάβισαρ ε, υπεγράμμισε ότι από το 2015 και μετά ο Διεθνής Οργανισμός ορίζει ότι μπορούν ε, τα πλοία που κινούνται στις περιοχές αυτές να χρησιμοποιούν καύσιμα με περιεκτικότητα κατά μέγιστο 1,5% σε θείο. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με προσπάθειες για τη βελτίωση του περιβάλλοντος. 0,5% που θα πρέπει τουλάχιστον στις συγκεκριμένε αυτές περιοχές να τηρηθεί από το 2012. Η συνέπεια ε, σε αύξηση κόστους θα είναι περίπου στο 40%, 60% εάν πρόκειται να τηρηθεί το ποσοστό του 0,1%. Για δε τα μεγάλα υπεροκειάνια ή μάλλον τα μεγάλα ποντοπόρα πλοία τα οποία θα πρέπει να διασχίζουν φερρυπίν τη μάχη για να περάσουν στο Τούρκο της Φινλανδίας για να μπορέσουν αυτά να διατηρήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ε, είναι σχεδόν ε, αδύνατο ή αδιανόητο με την ε, υποχρέωση για τήρηση των συγκεκριμένων ποσοστών. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι θα βρεθούν σε μειονεκτική θέση τα πλοία αυτά. Στην δε νότια όχθη της Μεσογείου προβλέπεται ένα ποσοστό 0,5%. Βεβαίως η πτυχή της υγείας, της δημόσιας υγείας έχει πολύ μεγάλη σημασία, πολύ σωστό αυτό, αλλά μην ξεχνάμε ότι η κατανομή, τουλάχιστον όπως βλέπω εγώ το κείμενο, για μένα είναι πολύ δύσκολο να γίνει κατανοητή. Δεν ξέρω εάν μπορώ να δεχθώ ανάλυση του τύπου τόσες χιλιάδες νεκροί στην Ευρώπη καφέτος λόγω της περιεκτικότητας εθίου. Σε θείο, αν θα είναι 10.000 ή 30, αυτό δεν μπορώ εγώ να το προβλέψω, ούτε να το, να το δεχθώ ως ανάλυση. Βλέπουμε ότι και ο Καναδάς και οι ΗΠΑ έχουν εισαγάγει τέτοιου είδους ε, περιοχές ελέγχου του θείου, στα 200 μίλια όμως, που δεν είναι δεσμευτικές ακόμη η δύναμοι των, των διατάξεων ε, του Διεθνούς Οργανισμού. Άρα, καλό θα ήταν να είμαστε πιο προσεκτικοί, να περιμένουμε, να δούμε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση και να διαφυλάσσουμε τις συνθήκες ανταγωνισμού για τις δικές μας ε, πλειοκτήριες εταιρείε, για την δική μας την ζώνη ε, βεβαίως να αποφύγουμε την μετακύληση από τις θαλάσσιες στις χερσαίες μεταφορές, γιατί μην ξεχνάμε ότι όταν λέγαμε ε, ε, ότι αντί να λέμε road to sea όπως λέγαμε άλλο αυτό το διάστημα, τώρα κινδυνεύουμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο του sea to road, να, με, να κυληθούν στις χερσαίες μεταφορές ε, τα φορτία αυτά. Και έτσι θα πρέπει να συζητήσουμε εάν Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Για το LNG, για το υγροποιημένο φυσικό αέριο βεβαίως, δεν έχω καμιά αντίρρηση. Θα πρέπει να υπάρχει όμως και αντίστοιχη δυνατότητα και υποδομή με δεξαμενές ε, ε, προμήθειας ε, σε υγροποιημένο φυσικό αέριο που να μπορεί να χρησιμοποιήσει το πλοίο. οι οποίες ακόμη δεν είναι έτοιμες. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η πρόθεση που αναφέρεται για το 2020, την εισαγωγή αυτών διατάξεων για το 2020 από το Διεθνή Αυτιλιακό Οργανισμό, μάλλον δεν θα είναι δυνατόν να τηρηθεί υπ' αυτές τις συνθήκες τουλάχιστον ακόμη. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Μέχρι 11 και 20 έχουμε χρόνο να σας υπενθυμίσω. Έχουν στήσει πολλοί συναδελφοί το λόγο. Πολλοί κυρίω από τι ε, βόρειε πλευρέ τη Ευρώπη και ο κύριο Κουμουτσάκο που ξέρω βεβαίω ότι έχει θεμητό ενδιαφέρον, αλλά πρώτα θα ακούσω τον κύριο Λιμπεράτσκι. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, την εισηγήτρια. Είναι σίγουρο ότι πρέπει να ασχοληθούμε με την οδηγία αυτή. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τις επιπτώσεις και όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά βεβαίως γνωρίζοντας ότι η οδηγία αυτή αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές, θα πρέπει να δούμε και τις επιπτώσεις που θα έχει όσον αφορά και τις δραστηριότητες των πλειοκτητών, αλλά και τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στους λιμένες. Διάβασα προσεκτικά όλα τα έγγραφα και θεωρώ ότι υπάρχουν πολλές δύσκολες και περίπλοκες πλευρές στο θέμα αυτό η, η συγγήτρια προετοίμασε μια ενδιαφέρουσα έκθεση. Το μεγαλύτερο τμήμα των προτάσεών της ε, μπορεί να με βρει σύμφωνο. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνούμε, λέγω, ότι η οδηγία αυτή δεν αφορά μονάχα τη Βόρεια Θάλασσα ή τις θάλασσες που είναι μόνο γύρω από τη Μάνχη. Αφορά και την Βαλτική Θάλασσα που είναι στην ουσία μια εσωτερική θάλασσα χωρών που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι η επίτευξη των ε, εν λόγω τιμών για το 2015 είναι ε, ε, αρκετά λογική η ημερομηνία. Τώρα, για τα πλοία τα οποία έρχονται έξω εκτός των χωρών ΣΕΚΑ, ναι, μπορεί να υπάρξει μια παρέκκληση για πέντε χρόνια. Μπορούμε να συμφωνήσουμε λοιπόν με αυτές τις προτάσεις και βεβαίως πιστεύω ότι θα πρέπει με μεγάλη προσοχή να ακούσουμε τις προτάσεις των πλειοκτητών γιατί καμιά φορά οι υπερβολικά εγωιστικές ε, προτάσεις ή υπερβολικές προτάσεις ε, μπορούν ακριβώς να μεταφέρουν ένα τμήμα των θαλάσσιων μεταφορών στις χερσαίες μεταφορές, στους δρόμους. Γενικώ πάντως συμφωνώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Βαντάλεν, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, κοιτάξτε, οι επικρίσεις ε, μπορεί να είναι πολυπληθείς ε, απέναντι στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός πήρε μια θεαματική κατά κάποιο τρόπο απόφαση. αλλά δεν ελήφθησαν υπόψη όλες οι επιπτώσεις και όλες οι πλευρές αυτής της απόφασης. Αυτοί που πήραν την απόφαση αυτή στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό ε, θα ε, έπρεπε να είχαν ε, υποβάλει κάποια εξαίρεση για μια επιπλέον χρονική ε, για ένα επιπλέον χρονικό περιθώριο. Ε, εγώ πιστεύω ότι οι θαλάσσιες μεταφορές πρέπει να γίνουν καθαρότητες, οπωσδήποτε θα πρέπει να γίνουν σεβαστές, ε, σεβαστά τα περιθώρια ή τα όρια των εκπομπών. Όμως, όμως, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι τα προβλήματα είναι πολλά. Ε, η διεθνή, ο Διεθνής Οργανισμός, οργανισμός πολλές φορές δεν λαμβάνει υπόψη της τις ε, επιπτώσεις που μπορούν ε, να υπάρξουν ε, μετά από μια τέτοιο είδους απόφαση και γι' αυτό και άλλωστε το αναφέρει και η συγκήτρια, ε, κινδυνεύουμε να έχουμε μεταφορά από τη θάλασσα ε, στους δρόμους των μεταφορών. Υπάρχει μάλιστα και μία μελέτη του Πανεπιστημίου της Λουβένης που ασχολείται ακριβώς με το θέμα αυτό και καταλήγει σε αυτό το ε, συμπέρασμα και ότι τελικά ε, με τέτοιες αποφάσεις θα καταφέρουμε απλώς να διονγκωθεί ακόμα περισσότερο ε, η, ο τομέας των χερσαίων μεταφορών όσον αφορά την μεταφορά εμπορευμάτων. Θα μπορούσατε λοιπόν να έρθετε σε επαφή με το Πανεπιστήμιο τη Λουβέννη, δεν ξέρω αν το έχετε κάνει ήδη. Θα ήταν ενδιαφέρον πάντω να μιλήσετε μαζί του. Ξέρετε κάτι, ο δρόμο για την κόλαση ε, είναι στρωμένο με καλέ προθέσει. Θέλουμε να κάνουμε κάτι καλό, αλλά εν προκειμένου, προσπαθώντα να κάνουμε ε, κάτι καλό, μπορεί τελικά να φτάσουμε σε ένα πάρα πολύ κακό αποτέλεσμα. Ε, θα πρέπει πραγματικά, ε, όταν γίνονται τέτοιε προτάσει, να έχουμε μια πολύ ακριβή ιδέα των αντικτύπων που θα έχει η απόφαση αυτή. Και εδώ δεν νομίζω ότι η ιδέα που έχουμε είναι πολύ σαφής. Θα έχουμε ε, στην ουσία, κατά την άποψή μου, ένα modal shift, ε, δηλαδή μετατόπιση των μεταφορών από τη θάλασσα στους δρόμους. Ε, υπάρχει επίσης και το συνολικό θέμα των καυσίμων 1,5-2% ε, εντάξει, όμως πιστεύω ότι η απόφαση προχωράει πάρα πολύ. Γιατί εδώ προβλέπεται τελικά απαγόρευση. Αυτό ήταν το δεύτερο μου. Τρίτον, θα πρέπει να ενδιαφερθούμε για τις εναλλακτικέ τεχνικές. Η εισηγήτρια έκανε κάποιο λόγο για το θέμα αυτό. Αναφέρθηκε στο θέμα αυτό. Για τα πλοία υπάρχουν τεχνικές καινούριες οι οποίες εμφανίζονται και υπάρχουν και εγκαταστάσεις οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα ε, να ε, καθαριστούν αυτές οι εκπομπές, οι πλυντηρίδες που λέμε και πιστεύω ότι οι πλειοκτήτες είναι έτοιμοι να επενδύσουν σε τέτοιες ε, καθαρές πολιτικές και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ πιο θετικό βήμα. Όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Και βεβαίως να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το ζήτημα της Βόρειας θάλασσας, της Βαλτικής θάλασσας και της Μάνχης. Εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρχει ομοιογενής πολιτική που θα εφαρμόζεται δηλαδή ταυτόσημα σε όλα τα ευρωπαϊκά ύδατα γιατί και η Μεσόγειος έχει ειδικά προβλήματα. Κατά την άποψή μου ε, θα πρέπει να ε, ε, έχουμε την ζώνη των 12 μιλίων έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί σε όλη την Ευρώπη γιατί διαφορετικά στη Μεσόγειο θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα. Ε, υποβάλλω λοιπόν το, το ζήτημα ε, αυτό. Μία ζώνη για όλη την Ευρώπη στα 12 μίλια. Ευχαριστώ πολύ Τέιλορ για τους ε, πράσινους. Um, Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ενδιαφέρουσα η συζήτηση, είναι πολύ καλό το σχέδιο και θα ήθελα να συγχαρώ τον συντάκτη, την συντάκτρια. Ακούγοντας τη συζήτηση μέχρι τώρα νομίζω ότι αυτό το οποίο θα δούμε είναι τα περί ποιότητας του αέρα. Έγιναν κάποιες συζητήσεις ε, για τους θανάτους, τον αριθμό των θανάτων που προκαλούνται από τις εκπομπές θείου. Και δεν νομίζω ότι μπορούμε να βάλουμε τιμή σε μια ζωή. Στηρίζουμε τη συμφωνία του Διεθνούς Ναυτιλικού Οργανισμού και αυτό πρέπει να αποτελέσει μια ακόμη σταθερά θα έλεγα. και θα πρέπει η σχετική νομοθεσία να περάσει στο ε, κοινοτικό ε, δίκαιο. Δεν νομίζω ότι πρέπει να καθυστερήσει η έγκριση, αλλά ούτε και η εφαρμογή. Άρα, ε, σε ό,τι αφορά τις προθεσμίες, συμφωνήσαμε ε, να παραταθεί η αξιολόγηση ό,τι αφορά τα αφαίρει, αλλά νομίζω ότι πρέπει να έχουμε την ίδια προθεσμία ε, με αυτή τη ΣΜΑΠΟ. Και σε ό,τι αφορά την προθεσμία του 2015 θα θέλαμε η αναβολή ως ε, ε, προθεσμία του 2025 με τις της πράξεις να διαγραφεί. Η... Τα επιχειρήματα για τη βελτίωση της πέτας του αέρα είναι τόσο συντριπτικά, είναι τόσο μαζικά, άρα νομίζω ότι θα πρέπει να επεκταθεί αυτή η διάταξη για τα χωρικά έδατα των κρατών μελών και θα έπρεπε και η Κομισιόν να κάνει την δέουσα ανάλυση. Και σε ό,τι αφορά κρατικές ενισχύσεις ε, για την εγκατάσταση ε, των συστημάτων καθαρισμού, ίσως ε, πάνω στα σκάφη, πάνω στα πλοία, αυτό θα έπρεπε ίσως να εξεταστεί. Και τώρα έρχομαι στο ίδιο το σχέδιο της έκθεσης. Νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρξουν ποιοτικά πρότυπα για τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στις ε, θαλάσσιες μεταφορές. Αυτό θα έπρεπε να το φροντίσει η Κομισιόν και επίσης οι έλεγχοι να επεκταθούν σε όλα τα ύδατα της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Να καλυφθεί όλη η ακτογραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, υπάρχουν και κάποια άλλα καινούρια θέματα τα οποία υπερβαίνουν το πεδίο εφαρμογή τη έκθεσης, τα οποία θα ήθελα να αναφέρω. Τα contaminated bunker fuels, όπως τα λέμε, πρέπει να συμπεριληφθούν. Και οι, οι διατάξεις της Marpol πρέπει να εφαρμοστούν πλήρως. Επίσης, ε, οικονομικά μέσα ε, ίσως είναι απαραίτητα για να λειτουργήσουν στην πράξη όλες αυτές οι διατάξεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, πρόεδρε, δεν είμαι, βέβαια, δεν έχω εμπειρία από τη ζωή των ναυτικών. Δεν είμαι ο ίδιος ναυτικός. Αλλά, εάν έχουμε καταφέρει να απαλλαγούμε ή να έχουμε καθαρά καύσιμα, καθαρό πετρέλαιο για τις οδικές μεταφορές, γιατί να μην το κάνουμε και για τις θαλάσσιες. Τώρα από την άλλη, αν θέλει ο καθένας να καίει ε, απόβλητα, τι να πω. Και όταν έχουμε καταφέρει να λύσουμε με την εισαγωγή της υποχρέωσης για, συγκεκριμένο, ε, για μια συγκεκριμένη απόσταση ε, να χρησιμοποιείται φυσικό αέριο για τις εναέρειες μεταφορές και έτσι έχουμε καταφέρει να καθαρίσουμε και τον αέρα των πόλεών μας γιατί να μην το κάνουμε και στις τελάσσες μεταφορές δεν θα είναι και αυτό δυνατόν Ίσως χρειαστεί να καλέσουμε μερικά ξωτικά ή κανένα άλλο κανένα νεραϊδοξωτικό να μας βοηθήσει και αυτό ίσως να είναι Άλλε αρχέ, όπως Φιλιππίνοι, Ηνωμένες και ο Καναδάς που έχουν εισαγάγει αυτό το όριο των 200 μιλίων. Και έτσι Αντίστοιχα, μπορούμε και στι ε, συνδιαλλαγέ μα και τι διαπραγματεύσει με τι χώρε τη νότια όχθη Μουσιογείου, για τι οποίε ακόμα δεν έχουμε καταλήξει, να συνεχίσουμε να επιμένουμε για να τι πιέζουμε να χρησιμοποιούν καύσιμα με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο. Εάν δεν τα καταφέρνουμε αυτά, ε, α σταματήσουμε πια να συνομιλούμε, α σταματήσουμε να μιλούμε για ολοκλήρηση και να σταματήσουμε να μιλούμε και για νέε προδιαγραφέ και όρια. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Ήκταλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και καταρχάς θα ήθελα να πω ότι έκανε πολύ καλή δουλειά η συγγετρία. Πολλές ε, εύστοχες παρατηρήσεις βλέπω στο κείμενό της, αλλά υπάρχουν ακόμα μερικά πράγματα που θα ήθελα να συζητήσουμε. Η πρόταση αυτή είναι μεγάλο πλήγμα για τον ε, κλάδο, ιδιαίτερα στις ε, βόρειες χώρες. Κατά μια χρονική στιγμή κατά την οποία χρειάζεται περισσότερη υποστήριξη εθνικής οικονομίας, φοβούμε ότι αυτή η νέα τεχνολογία δεν ε, θα είναι δυνατόν να ε, εισαχθεί κατά τρόπο ανώδυνο και για να τηρηθεί βέβαια το όριο που προβλέπεται. Και επίσης ανησυχώ για το γεγονός ότι έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα toolbox, ε, μια εργαλειοθήκη για τη στήριξη των κρατών που θα πληγούν από τα νέα όρια. Θα ήθελα πολύ πιο σαφείς διατυπώσεις για το πώς θα μπορούσε ο ναυτιλιακός κλάδος οικονομικά και βιώσιμο να τηρήσει αυτές τις ε, υποχρεώσεις της μεταβατικής περίοδου. Επίσης, η δυνατότητα που αναφέρεται ήδη στην έκθεση χάσει για την επέκταση των περιορισμών στο 0,1% ε, σε περιοκταθείου για τις στρατιωτικές χρήσεις, τα στρατιωτικά απλή, έτσι ώστε να εξασφαλιστούν ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Θα ήθελα να δω τι μοίρα έχει. Ευχαριστώ κύριε Σκουμουτσάκος. Ευχαριστώ ε, κύριε Πρόεδρε. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι η έκθεση είναι μια καλή βάση για συζήτηση και θα υπάρξουν, ε, είμαι σίγουρος, ε, διάφορες σκέψεις και τροπολογίες πάνω σε αυτές. από εκεί και πέρα παίρνω τη συνέχεια από αυτό που μόλις ακούστηκε από τον συνάδελφο τον κύριο Ιταλά. δεν θα πρέπει να προχωρήσουμε τόσο πολύ ώστε τελικά να φέρουμε το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Να επιβαρύνουμε τις χερσαίες μεταφορές και ουσιαστικά να καταλήξουμε σε μια επιβάρηση του περιβάλλοντος με μια λαθασμένη πολιτική που δεν θα λύνει τίποτα, θα δημιουργεί πρόβλημα στην ανταγωνιστικότητα του ναυτιλιακού τομέα και επιβάρηση του περιβάλλοντος γιατί θα έχουμε μετακίνηση στις χερσαίες μεταφορές. Ε, επομένως θα πρέπει να αναζητήσουμε και εδώ μια ισορροπία, μια λεπτή ισορροπία η οποία είναι εφικτή. Ε, ίσως το 2015 είναι μια ημερομηνία που δεν νομίζω ότι είναι ρεαλιστική. Θα πρέπει να κινηθούμε πέραν του 2015 και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας αυτό και το γεγονός ότι ε, μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα που μένει πολλά από τα λιμάνια ε, στην Ευρώπη δεν θα έχουν τη δυνατότητα τις εγκαταστάσεις αλλά και τις τεχνικές δυνατότητες να προμηθεύουν αυτό το ειδικό καύσιμο. Πράγμα το οποίο ε, σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να ζητάμε από τα πλοία που θα, επιβεβαιώ, θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την ανταγωνιστικότητά τους να αλλάζουν πορεία για να πηγαίνουν σε άλλα λιμάνια που έχουν αυτό το καύσιμο. Βλέπουμε λοιπόν, αυτό το ανέφερα, μόνο σε ένα από τα τεχνικά προβλήματα που έχει η εφαρμογή αυτή. Λοιπόν, κλείνοντα, θέλω να πω ότι ναι, μεν κινείται σε σωστή κατεύθυνση ε, το κείμενο που συζητάμε, αλλά θα πρέπει να γίνουν ορισμένε διορθώσει για να γίνει πιο ρεαλιστικό και τελικά πιο αποδοτικό για τον τελικό του σκοπό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Φλάκενστάιν. Πρόεδρε, όπως έχει κατάσταση σας προς τη ρήπαρση του περιβάλλοντος από τα πλοία, διαπιστώνουμε ότι πολύ λίγα πράγματα έχουν γίνει μέχρι τώρα και ότι θα πρέπει πλέον να αλλάξουμε αρκετά πράγματα στις εκπομπές. Πρώτον, αυτό είναι σαφέ, νομίζω για όλου. Δεν υπάρχει αντίρρηση. Άλλωστε το έχουμε αποφασίσει, το έχει πει και ο διεθνή Αυτοκρατικό οργανισμό. είναι ο Στόχο. Δεύτερον, δεν βλέπω γιατί θα πρέπει μόνο στα βόρεια, στις βόρειες ακτές Ευρωπαϊκής Ένωσης να, εισάγουμε, να εισαχθούν τέτοιου είδους όρια. Και σε τελευταία ανάλυση θα πρέπει να φροντίζουμε και για τη δημόσια υγεία και στη Νότια Ευρώπη. Γιατί θέλουμε να προστατεύσουμε μόνο τους ε, Ευρωπαίους του Βορρά Ακούσαμε βέβαια τα αριθμητικά που μας αναφέρατε, αλλά τους άλλους του Νότου τους αφήνουμε στη μοίρα τους. Τρίτον, ο κύριος Φαντάλεν βεβαίως και έχει δίκαιο ότι δηλαδή θα πρέπει να προβλεφθούν ισοσκελιστικά μέτρα, ισοσκελιστικές λύσεις εξ αρχής, έτσι ώστε να μην πληγεί κανείς κατά τρόπο ανισομερή. Και πιστεύω ότι θα θυμάστε κι εσείς πως είχαμε ζητήσει μια μελέτη σχετική, αλλά δεν τη βλέπω πουθενά. Έχει γίνει αυτή η μελέτη, δόθηκαν κάποιες απαντήσεις. Για δε την ασφάλεια. Δεν ξέρω επίση αν έχουν προχωρήσει οι μελέτες ε, στο θέμα αυτό, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει αρκετή πρόοδος. Και ίσως θα χρειαστεί μια φάση, μια περίοδος σταδιακής εισαγωγής, phase in δηλαδή των μέτρων Κατά τα άλλα όμως θεωρώ ότι ο βασικός στόχος πρέπει να τηρηθεί με αυτές τις εξαιρέσεις, τις Ευχαριστώ κύριε Φλέκενστάιν. Είχαμε όντως αναθέσει σε έναν αντισυμβαλόμενο τη μελέτη, αλλά ο αρχικός ανάδοχος απεσύρθη εν τέλει και γι' αυτό δεν την έχουμε. Πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να την έχουμε εγκαίρως για να ληφθεί υπόψη. Όπως ήθελα να υπογραμμίσω όμως, ε, δεν την έχουμε μέχρι τώρα διότι απεσύρθη ο ανάδοχος. Ο κύριος Κράμερ έχει το λόγο. Μπορώ να συμφωνήσω με τον κύριο Φλέκενστάιν για τις τρεις πρώτες του παρατηρήσεις και βεβαίως πάντοτε λέγαμε ότι ε, περιμένουμε να ακούσουμε πάντα ότι ε, πάντα ακολουθούσε ο Διεθνής Αυθυλιακός Οργανισμός τα όσα είχαμε εμείς να πούμε ε, στα όσα διεκδικούσαμε εμεί. Και τώρα, μία φορά που έρχεται ο Διεθνή Αυτιλιακό Οργανισμό να ζητήσει μια, φορα που ερχεται ο Διεθνής Αυθυλιακός Οργανισμός να ζητησει μια μια λύση και μέτρα, εμεί προσπαθούμε να τραβήξουμε το φρένο. Ε, δεν γίνεται λοιπόν. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι δεν έχουμε να κάνουμε με κάψιμα απόβλητα και με απόβλητα. Περί αυτού πρόκειται. Μολύνουμε το περιβάλλον, καταστρέφουμε τη ζωή. Και θα ήθελα να πω ότι η σύγκριση με τη Μεσόγειο βεβαίω μπορεί να ισχύει, αλλά κάντε μία προσπάθεια να δείτε πού βρίσκονται και οι σχετικές εκστρατείε ενημέρωσης και διαφήμισης. Έχετε δει καμιά εκστρατεία διαφημιστική για τις χώρες του Βορρά η οποία θα καλούσε τους τουρίστες αντί να πηγαίνουν στις μεσογειακές ακτές να έρθουν στις χώρες του Βορρά και να πούνε και εμείς έχουμε θάλασσες και εμείς έχουμε παραλίες και μάλιστα έχουμε και καθαρό περιβάλλον και μην πηγαίνετε στην νότια, στην νότια Ευρώπη, στη Μεσόγειο δηλαδή γιατί εκεί είναι ε, μολυσμένα τα νερά, μολυσμένος ο αέρας και θα αρρωστήσετε και θα πεθάνετε αν πάτε στις χώρες αυτές. Αυτό θέλετε να γίνετε. Μπορούμε να το κάνουμε. Πρέπει να σκεφτούμε δηλαδή ότι η Βαλτική δεν είναι μια θάλασσα η οποία προορίζεται μόνο για, την, για τις θαλάσσιες μεταφορές. Δεν είναι δηλαδή μονοπόλιο των πλοίων. Είναι ένας παράδεισος για τον τουρίστα, για τον επισκέπτη. Αν αναλογιστούμε δε τι είδου συνέπειε μπορεί να έχει η ρήπανση του περιβάλλοντο οικονομικά, τα 15% τη προσαρμογή που αναφέρατε είναι ψίχουλα. Παραλαμβάνω, οι εσωτερικέ θαλάσσιες μεταφορέ είναι οικολογικέ, είναι φιλοπεριβαλλοντικέ, μόνο εφόσον τηρηθούν συγκεκριμένα όρια στι εκπομπέ. Και βεβαίω. Εδώ θα πρέπει να σημειώσω ότι διαφοροποιούμαστε σε σχέση με τις μικρομεσαίες ή τις μεγάλες επιχειρήσεις. Οι μεγάλες επιχειρήσεις βεβαίως μπορούν να πληρώσουν και αυτό το ποσό και το τριπλάσιο του ποσού. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έχουν τη δυσκολία. Χαίρομαι λοιπόν που ιδιαίτερος υπό αυτές τις συνθήκες η Διεθνής Ναυτιλιακή Οργάνωση ήταν εκείνη η οποία έλαβε την απόφαση και άρα μπορεί να επιβάλλει και τις κυρώσεις στους λιμένες εκείνους οι οποίοι δεν τηρούν τις προδιαγραφές διότι δεν είναι δυνατόν αυτοί που προσαρμόστηκαν εγκαίρως να βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση και εκείνοι που είπαν «Α, τώρα σιγά μην προσαρμοστούμε, σιγά μην, μην κάνουμε αυτό που ζητούν οι κυβερνήσεις» και έχουν απλώς χρονοτριβήσει, να επωφελούνται από ε, το γεγονός αυτό και μόνο, το δηλαδή ότι δεν είναι έτοιμοι. Έχουμε πάντοτε εισαγάγει μέτρα δύσκολα που έγιναν αποδεκτά όταν μπορούσαμε με ισχυρή πολιτική βούληση να τα στηρίξουμε και το ίδιο πράγμα νομίζω μπορεί και πρέπει να γίνει και στον τομέα των θεράσεων μεταφορών. Ο κύριος Βίμπερ από την Επιτροπή. Θέλετε να μιλήσετε. Α, όχι, κύριε Μάιτζεν πρώτα. Όχι. Δεν σας είχα γραμμένη στον ε, καταλογό μου, αλλά βεβαίως σας δίνω το λόγο. Ναι, νόμιζα ότι έρχεται η σειρά μου, γι' αυτό δεν ζήτησα το λόγο. Ε, είναι ένα θέμα το οποίο με έχει απασχολήσει εδώ και πολύ καιρό. Ο Διεθνή Αυτιλιακό Οργανισμό είναι προφανώ ότι δεν θα πρέπει να τροποποιηθεί. Αυτό είναι βέβαιο, γιατί πρόκειται για μια απόφαση που έχει ληφθεί σε παγκόσμιο επίπεδο και όχι σε ευρωπαϊκό. Βεβαίω θα πρέπει να δούμε το κατά πόσο μπορεί να υπάρξει αναβολή. Υπάρχει αναβολή για τι περιοχέ εκείνε που βρίσκονται έξω από τα ΠΕΘ Άλλες περιοχές μπορούν να τηρήσουν ε, την ε, χρονική περίοδο του 2015, άλλοι το 2020 θα πρέπει να είναι στο 0,5%. Κανονικά δεν προβλέπεται δηλαδή αναβολή, ίσως θα μπορούσαμε να τη συζητήσουμε. Για την ε, δε έκθεσή μου για την ολοκληρωμένη πολιτική για τι θάλασσε, έχω συμπεριλάβει δύο παρατηρήσει που είχαν να κάνουν με τις καθαρές θάλασσες, θάλασσε μεταφορέ. Το ένα ότι χρειάζεται μια υποστήριξη οικονομικού χαρακτήρα για την οικολογική θαλάσσια μεταφορά, για τι οικολογικές θαλάσσιες μεταφορέ. Κάποιοι είπαν ε, μάλιστα ότι υπάρχουν ήδη πράσινα πλοία, ναυπηγούνται σε ορισμένες περιοχές, να, πράσινα πλοία και σε κάποιες άλλες, σε κάποια άλλα ναυπηγεία όχι και άρα θα πρέπει να δοθεί μια προτίμηση και να προωθηθούν τα πιο οικολογικά πλοία και βεβαίω το θέμα των εκπομπών στη Βόρεια και τη διαφοροποίηση με την Νότια Ευρώπη είχα αναφέρει. Υπάρχει ο κίνδυνος, λέτε, ότι μπορεί να μετακυλιστεί η, ε, το, το φορτίο από τις θαλάσσες στις χεσές μεταφορές. Αυτό δεν είμαι βέβαιη ότι μπορεί να συμβεί. Ε, υπάρχουν δηλαδή μελέτε που δείχνουν το αντίθετο, την αντίθετη εξέλιξη, την αντίστροφη εξέλιξη. Βέβαια, αυτό δεν θα πρέπει να το επιτρέψουμε όπω και να έχει. Θα πρέπει δηλαδή να φροντίσουμε να αποτρέψουμε, να ένα τέτοιο κίνδυνο. Υπάρχουν διάφορε. Ε, διαδικασίες, ξηρή διαδικασία ή υγρή ε, διαδικασία ε, για την σύλληψη του θείου, η οποία στην, ξηρή, ε, στην υγρή διαδικασία ουσιαστικά τα πάντα εκλείονται μέσα στη θάλασσα, απελευθερώνονται μέσα στη θάλασσα και φυσικά αυτό προξένει τη μεγάλη ρήπανση. Και άρα δεν το προτιμούμε, προτιμούμε την ξηρή διαδικασία σύλληψη, η οποία σχεδόν μέσα σε αλίδια μπορεί να, να, να συλλάβει και να κρατήσει το θείο. Επίση η ανάμειξη με το υγροποιημένο φυσικό αέριο, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι έχουμε ένα σεμινάριο την επόμενη εβδομάδα για το πώ το υγροποιημένο φυσικό αέριο μπορεί να αποτελέσει ένα ε, μια εναλλακτική λύση. Είναι μια καλή πρόταση και πιστεύω ότι χρειάζεται η προσαρμογή των τεχνικών ε, υποδομών, των, των εξοπλισμών δηλαδή. Επίσης θα ήθελα να αναφέρω και την ε, αναφορά της εισηγήτριας ε, στις ε, παρεμβατικέ μεταφορές στην Νότια Ευρώπη ε, περίμενα να έχω περισσότερε αντιδράσεις από τους συναδέλφους στις προτάσεις συγκήτρια, περισσότερες από ό,τι είδα τελικά, αλλά νομίζω ότι έχει δίκιο. Δηλαδή, οι εκπομπές διοξιδίου του θείου είναι ρηπογόνος παράγοντας, σημαντικός για την ατμόσφαιρα και άρα θα πρέπει να αποτρέπεται. Ευχαριστώ η Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Χαιρετίζει η Κομισιόν το σχέδιο έκτασης και ευχαριστεί και την εισηγητρία για το έργο και την ε, στήριξη που ε, δίνει στην πρόταση. Θα θέλαμε να αναφερθούμε σε κάποια από τα θέματα τα οποία αναφέρθηκαν και πρώτα απ' όλα σε ό,τι αφορά τις εκπομπές από τα πλοία. Να το βάλουμε αυτό το θέμα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Πόρο απέχουμε του να πετύχουμε τους περιβαλλοντικούς μας ε, στόχους δηλαδή να μην έχουμε επιδείνωση της ποιότητας του αέρα που θα επηρεάσει αρνητικά και θα θέσει σε κίνδυνο τόσο το περιβάλλον όσο και την ανθρώπινη υγεία. Ο περιβάλλον αέρα σε κάποιες παράκτιες πόλεις ε, ο ατμοσφαιρικός αέρας θα ε, ρηπανθεί πολύ σημαντικά από τις ε, ε, εκπομπές ε, καυσαριών από τα πλοία και είναι πάρα πολλά τα βαρέμετα σωματίδια τα οποία αναπνέει ο κόσμος. Ε, στη Σικελία για παράδειγμα μεγάλη ατμοσφαιρική ρήπανση που προέρχεται από τα πλοία. Προσπαθούμε να περιορίσουμε ιδίως τις εκπομπές διοξιδίου του θείου που μετατρέπεται σε συγκεκριμένα μέταλλα και είναι ένας ρήπος που επηρεάζει πάρα πολύ ε, αρνητικά την ανθρώπινη υγεία και έχουμε κάνει ε, κάποια επιτυχία σε αυτές τις προσπάθειες. Τώρα, το θέμα των εκπομπών από την ακτοπλοεία, από τα πλοία είναι ε, κάτι που το οποίο θα μας επιτρέψει να καταπολεμήσουμε πολύ αποφασιστικά τις εκπομπές διοξιδίου του θείου. Οι περισσότερες χώρες δυσκολεύονται να εκπληρώσουν τα απαραίτητα πρότυπα, αλλά με το στόχο, με το εργαλείο αυτό είναι ένας πολύ φθηνός τρόπος για να τα καταφέρουν. Μετά από πολλά χρόνια που δεν είχαμε καλή νομοθεσία, πλέον βλέπουμε ότι έχει έρθει σειρά και του ε, ναυτιλιακού τομέα. Πρέπει και τα πλοία να συνεισφέρουν. Στη Βόρεια Ευρώπη έχουμε τους, ε, τις προχές ελέγχου ε, για τις εκπομπές ε, θείου και αυτό γίνεται από περιβαλλοντικές παραμέτρους. Έχουμε πρόβλημα στη Βόρεια Ευρώπη γιατί τα οικοσυστήματα είναι πιο ευάλωτα εκεί. Οι περιοχές αυτές λοιπόν ε, είναι και οι σκαπανείς αν θέλετε, οι πρωτοπόροι στην προσπάθεια αυτή. Η Κομισιόν ε, επικεντρώνεται στην, ε, στον αντίκτυπο για την υγεία. Έχουμε περιπτώσεις που έχουμε κάποια τέτοια περιοχές ελέγχου και στην Νότια Ευρώπη επειδή το ζήτησαν τα κράτη, τα συγκεκριμένα. Αλλά αυτό που θέλουμε είναι μια πρόταση που ε, θα στηρίζεται από όλα τα κράτη ε, να γίνει η ΣΕΚΑ, ε, η Βαλτική, η Βόρεια Θάλασσα. Αλλά υπάρχουν θάλασσες όπως η Μεσόγειος, παραδείγματο χάρη, ή το Ιρλανδικό Πέλαγος που δεν είναι ακόμα ΣΕΚΑ, δηλαδή περιοχές ελέγχου εκπομπών θεού γιατί δεν έχει ζητηθεί αυτό από τα κράτη-μέλη. Εμείς θα αξιολογήσουμε την σκοπιμότητα, το κόστος, το όφελος της κήρυξης επιπλέον θαλάσσιων περιοχών ως περιοχών ελέγχου εκπομπών στο πλαίσιο της πολιτικής και της αναθεώρησης πολιτικής για την ποιότητα του αέρα. Έχουμε δρομολογήσει και μία μελέτη, η οποία θα επικαιροποιήσει τα στοιχεία για τις εκπομπές ε, θείου και θα δούμε τα διάφορα σενάρια. Αν ε, μειωθούν διάφορες εκπομπές ε, και να δούμε αν θα μπορούσαμε να βρούμε και κάποιες άλλες θαλάσσιες περιοχές που θα υπήρχε πραγματικά καθαρό όφελος αν αυτές οι περιοχές ορίζονταν ως περιοχές ελέγχου εκπομπών. Βέβαια, δεν υπάρχει λόγος να καθυστερήσει η προβλεπόμενη εισαγωγή των απαιτήσεων σε ό,τι αφορά το θείο ε, στις βόρειες περιοχές ελέγχου εκπομπών. Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχουν κάποιες διατάξεις ε, για τη μείωση των ε, εκπομπών από τα πλοία που θα έχει τρομερό αντίκτυπο. Για κάθε ευρώ το οποίο επενδύουμε θα έχουμε 25 ευρώ όφελος. 25 ευρώ κέρδος. Το 90% περίπου ε, των ε, επιδομάτων υγείας, ε, ασθενείας, είναι σε χώρες που είναι κοντά σε περιοχές ελέγχου εκπομπών. Και αν θέλετε να σας δώσω και συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία για να έχετε κάτι έτσι πιο απτό στα χέρια σας, οι διατάξεις ΕΚΑ αποτρέπουν τον πρόωρο θάνατο 23 βρεφών. 16.000 ενηλίκων ετησίως επίσης. Άρα, εάν υπάρξει καθυστέρηση στην εισαγωγή αυτών των διατάξεων, θα ε, πεθάνουν προώρα 100 παιδιά και σχεδόν 19.000 ε, ενήλικοι. Ε, με την οικονομική κρίση που υπάρχει μπορούμε να δεχθούμε τέτοιες απώλειες σε ανθρώπινο κεφάλαιο. Ε, η Κομισιόν τώρα αντιμετωπίζει τα διάφορα ζητήματα που έχουν προκύψει. Έχουμε αναθέσει μελέτες και έχουμε ζητήσει και από τον ε, Οργανισμό Ασφάλειας ε, των Θαλάσσιων Μεταφορών να μας πει ε, ποιος είναι ο κοινό παρονομαστής των όλων μελετών. Από τα όλα στοιχεία προέκυψε ότι η εισαγωγή των νέων καυσίμων, ο ε, θα έχουμε αύξηση μένει στις τιμές ε, των καυσίμων. Άρα αυτό μπορεί να επηρεάσει το υπόδειγμα των μεταφορών, αλλά για να τα πω έτσι πιο συνεκτικά, το συμπέρασμα είναι ότι θα επηρεαστεί μεν το μέσα εκτοπλές, αλλά δεν περιμένουμε μείωση στα ε, σύστημα των εμπορευματευτικών μεταφορών. Ίσως μειωθεί το μερίδιο στην ανάπτυξη του κλάδου, γιατί μιλάμε για ε, στοιχεία 2,9 για τις εμπορευματικές και 3,5 για τις επιβατικές μεταφορές. Ίσως υπάρξουν ε, σε κάποιες διαδρομές, ε, σε κάποιες γραμμές περιορισμοί και η Κομισιό θα παρακολουθεί τις εξελίξεις εκ του ε, στον τομέα αυτό για να δει κατά πόσον θα πρέπει να αντιδράσει με κάποια μέτρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη θεσιμότητα των καυσίμων, ένα θέμα το οποίο ετέθη, η Κομισιόν θεωρεί ότι η διαθεσιμότητα των καυσίμων δεν είναι και τόσο μείζον ζήτημα τα καύσιμα ΣΕΚΑ αντιστοιχούν σε ένα μικρό μερίδιο σε σχέση με τα συνολικά θαλάσσια καύσιμα. Επομένω, μιλάμε για λίγε ποσοστίε μονάδε. Προβλέπουμε λοιπόν ότι θα υπάρχουν διαθέσιμα καύσιμα. Όμω από την άλλη πλευρά, σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμα καύσιμα, υπάρχει η τρέχουσα εκδοχή ε, της οδηγίας που προβλέπει μία ρήτρα παρέκκληση σε περίπτωση μη διαθεσιμότητα. Τα κράτη-μέλη κοινοποιούν λοιπόν στην Κομισιόν και έτσι μπορεί να ανασταλεί η ε, ισχύουσα απέτηση για τα καύσιμα. Υπάρχει ήδη μια σχετική διάταξη λοιπόν και πολλοί εμπλεκόμενοι φορείς έχουν ζητήσει την εισαγωγή αυτής της ρήτας μη διαθεσιμότητας που έχει αναπτύξει ο Διεθνής Αυθυλιακός Οργανισμός και την εισαγωγή της στην οδηγία. Σε ό,τι αφορά ε, την τεχνολογία scrapping υπάρχουν ε, ε, διάφορες απόψεις. Εμείς θεωρούμε ότι για να μπορέσει να τηρηθεί η απέτηση του Διεθνούς Αυθυλιακού Οργανισμού σε θέση με το θέμα αυτό, Νομίζουμε ότι θα πρέπει να εγκριθούν τα μέτρα έγκαιρα, πρόωρα. Εδώ είναι ανοιχτό το θέμα των ε, κρατικών ενισχύσεων. Μην περιμένετε άμεσε ενισχύσει από την Κομισιόν βέβαια. Αλλά επιτρέπονται κρατικέ ενισχύσει για όσου ε, υπερβαίνουν τα περιβαλλοντικά πρότυπα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δηλαδή εισαγάγουν ε, τα μέτρα νωρίτερα ή αν υπερβούν, αν έχουν ακόμη πιο αυστηρά πρότυπα και μέτρα σε ισχύ. Η Κομισιόν ελπίζει να μην ξαναδιδαχθούμε κάποια ε, διδάγματα αρνητικά. Υπήρχε μια μεγάλη καθυστέρηση στην ε, εφαρμογή κάποιων μέτρων. Εμείς θέλουμε λοιπόν η να υπάρχει έγκαιρη έγκριση της σχετικής διάταξης. Δεν ξέρω αν θέλει η κάτι να προσθέσει. Ε, ναι, ευχαριστώ. Θα ήθελα σύντομα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς τους συναδέλφους που έλαβαν το λόγο. Όντως, όλα αυτά τα θέματα τα συζητήσαμε με τους ενδιαφερόμενους φορείς. Θα ήθελα να υπογραμμίσω η κύρια έκθεση ανήκει στην, ε, η έκθεση ανήκει στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ορισμένες από τις έννοιες δηλαδή ε, φερειπίν ε, περιεκτικότητα σε οξύδια του, σε του αζότου και ε, το ζήτημα του χαρακτηρισμού της ρήπανσης έχουν ήδη κρυφθεί από την Επιτροπή Περιβάλλοντος και δεν ε, μας αφορούν εμάς. Εγώ προσπάθησα να δω μόνο τις πτυχές που έχουν να κάνουν με την δική μας Επιτροπή, με τις μεταφορές δηλαδή, αν και βέβαια μέλημα των πάντων είναι πάνω απ' όλα η προστασία του περιβάλλοντος και βεβαίως με ε, μέτρα όπως τα 200 μιλιά Ε, θα πρέπει να δούμε πώς θα το χειριστούμε, διότι υπάρχουν υποχρεώσεις που νομικά μας δεσμεύουν από την αρχή της ε, λειτουργίας συμφωνίας. Δεν μπορούμε δηλαδή να αναβάλουμε την εφαρμογή της συμφωνίας, εκτός και αν κάποιες επιχειρήσεις για ορισμένους τομείς ε, δείξουν την διάθεση να αν ε, προσαρμόσουν τις εργασίες τους, όπου θα μπορούσαμε να δώσουμε ένα περιθώριο έτσι ώστε να μην βρεθούν σε μειονεκτική θέση, να μην ε, αντιμετωπίσουν ε, μέτρα δυσμένη. Θα ήθελα επίση να επισημάνω ότι μπορεί να έχουμε διαφορετική μεταχείριση προ τι ε, μικρέ αποστάσει και τι μεγάλε αποστάσει, όπω αντίστοιχα έχουμε την Ευρωβινιέτα στα φορτηγά. Θα μπορούσαμε να εισαγάγουμε ένα σύστημα για τι τεράστιε μεταφορέ μεγάλων αποστάσεων. Φυσικά, ε, ευχαριστώ τους πάντες για τη συμμετοχή τους στη συζήτηση και κάποιες από τις τοπολογίες θα πρέπει να τις προσαρμοστούν για να καταστεί πιο σαφές ε, το κείμενο. Η κυρία Φώστερ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να καταστεί σαφέ το εξή. Βέβαια, όλοι μα θέλουμε να σημαίνουμε το δυνατόν πιο καθαρό περιβάλλον και θα ήθελα να επισημάνω το εξή και να διαφοροποιηθώ, γιατί βεβαίω έχει το δικαίωμα η συγγήτρια να ε, διατυπώσει ό,τι προτάσει θέλει, ένα δικαίωμά τη, όπω είναι και τη Επιτροπή, να διατυπώσει τι θέσει. Αλλά ρωτώ, 17.000 νεκροί που μου λέτε, πού το βρήκατε, πώ το, αποθεί, πώς το αποδεικνύεται, τα δεν ξέρω πόσε εκατοντάδες πρόωρα νεοχνά Πού το βρήκατε, πώς έχει αποδειχθεί αυτό. Εγώ έχω μεγαλώσει σε λιμάνι, ε, έχω γεννηθεί και μεγαλώσει σε λιμάνι, ζω σε λιμάνι καθημερινά, επομένως μου φαίνεται πολύ δύσκολο να δίνετε τόσο αυστηρούς και ακριβείς ορισμούς ή ε, αριθμούς καλύτερα για τις συνέπειες της χρήσης του θείου στα καύσιμα δεν χρειάζεται λοιπόν να μας παίρνετε όλους για ανόητους, δεν είμαστε ανόητοι και δεν χρειάζεται να μας φοβίζετε με κάποιο ε, ανδρίκελο, με κάποια, με κάποια νούμερα ε, τρομακτικά για να μας υποχρεώσετε να λάβουμε αποφάσεις. Ευχαριστώ λέει ο ψηφίσουμε το θέμα, εξετάζουμε το θέμα αυτό πάλι τον Νοέμβριο, ψηφοφορία το Δεκέμβριο και Επιτροπή Περιβάλλοντος, ε, από ό,τι κατάλαβα, το βλέπει τον Γενάρη. Και τώρα το επόμενο θέμα στην ημερησία διάταξη είναι η παρουσίαση της οδηγίας ε, για την, ε, των οικονομικών πτυχών καλύτερα της βιώσιμης κινητικότητας. Παρουσίαση μελέτης. Ο κύριος Wolfgang Schade και ο κύριος Werner Rottengatter είναι εδώ παρόντες για να μας παρουσιάσουν τη μελέτη τους. So we have about 20 minutes to... 20 λεπτά έχετε στη θέση σας για την παρουσίαση. Για να έχουμε ένα μικρό περιθώριο μετά για ερωταποκρίσεις. περίπου 15 λεπτά. Έτσι ώστε να τελειώνουμε το μεσημέρι τη συνεδρίαση. Γιατί κουραστήκαμε πιστεύω όλοι με τις ψηφοφορίες και κυρίως από το γεγονός ότι το τσάι μας ξέχασε και δεν μας ήρθε. Ποιος θα αναλάβει λοιπόν πρώτος. Ο Δόκτωρ Σάντε, ο κύριος Ρότενμπεργκερ, ο κύριος Σάντε. από την Gesellschaft Fraunhofer, δεν ξέρω αν τα γερμανικά μου αρκούν για να καταλάβετε τι θέλω να πω, από το Ινστιτούτο Fraunhofer λοιπόν και ο κύριος Ρότιν Κάτερ είναι από το Ινστιτούτο της Καλσρουής, ε, τεχνολογικό το Καλσρουής, αυτό τουλάχιστον μπορώ να το προφέρω. Ευχαριστώ, έχετε το λόγο. Okay. Thank Ευχαριστώ πολύ Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα της μελέτης μας για τις οικονομικές πτυχές της βιώσιμης κινητικότητας. Είναι μια κοινή παρουσίαση που θα γίνει μεταξύ μου και του συναδέλφου του κύριου Ρότεν Γκάτερ. Ο σας ε, ε, είπε τα σχετικά. Μας έχει ήδη συστήσει. Ε, θα σας μιλήσω λοιπόν ε, για την ε, μελέτη, πώς συγκροτήθηκε, το αναλυτικό πλαίσιο επίσης. Δεν μπορούμε μέσα στα 20-25 λεπτά να σας πούμε όλες τις λεπτομέρειες, αλλά μπορείτε να διαβάσετε τα σχετικά. Και έπειτα θα αναφερθώ σε κάποια συμπεράσματα και εν τέλει στις υποδείξεις και συστάσεις που διατυπώνονται στη μελέτη. Λοιπόν, η μελέτη μας. Ε, καθορίσαμε πρώτα απ' όλα τους όρους, κάποιους πολύ ε, σημαντικούς όρους για να ορίσουμε την οικολογική καινοτομία η οποία προωθεί την ε, βιώσιμη κινητικότητα. Πέντε στοιχεία βασικά και με βάση αυτά αναπτύξαμε έναν πολύ μακρύ κατάλογο πολιτικών καινοτομίας, 8-9 καινοτομίες συγκεκριμένα, των οποίων χρησιμοποίησαμε ένα αναλυτικό πλαίσιο για να καταλήξουμε σε ένα πιο σύντομο κατάλογο των ε, σημαντικότερων οικολογικών καινοτομιών κινητικότητας. Και μετά κάναμε μία πλήρη ανάλυση με τη βοήθεια αυτού του αναλυτικού πλαισίου. Εκ παραλλήλου κάναμε και μία online έρευνα για να συμπληρώσουμε τα πορίσματά μας ε, για τις ε, οικολογικές αυτές καινοτομίες. Με όλες αυτές τις δραστηριότητες ε, συναγάγαμε και τα συμπεράσματα μας καθώς και τις συστάσεις μας οι οποίες αφορούν τις οικονομικές πτυχές της βιώσιμης κινητικότητας. Ποιε ήταν οι υποθέσει μα, ε, τι κατανοούμε λοιπόν με του όρου ε, πρώτα απ' όλα βιώσιμη κινητικότητα. Δεν μιλάμε μόνο για τι μεταφορικέ δραστηριότητε, μιλάμε και για την προσβασιμότητα, τη προσπελασιμότητα, τι δυνατότητε που παρέχει το σύστημα των μεταφορών στου χρήστε. Και δεύτερο, στοιχείο το οποίο θα πρέπει να αναφέρουμε εδώ είναι ότι βέβαια θεωρούμε ότι και οι τρει διαστάσει τη ε, βιωσιμότητα, οικολογική, περιβαλλοντική, κοινωνική, λαμβάνονται υπόψη. Έτσι εννοούμε εμεί λοιπόν την βιώσιμη κινητικότητα στη μελέτη. Δεύτερο σημαντικό όρο όρος. Eco-innovation, οικολογική καινοτομία. Τι είναι λοιπόν ένα καινοτόμο μέτρο. Είναι ένα μέτρο το οποίο θα πρέπει τουλάχιστον να, οδηγεί σε κάποια περιβαλλοντική βελτίωση όταν εφαρμόστε δηλαδή αυτή την επίπτωση να έχει. Και βέβαια δεν θα πρέπει να είναι η προτεραιότητα ε, το πώς υλοποιών, ε, γιατί υλοποιείται. Θα μπορεί να υλοποιείται για τη βελτίωση της αποδοτικότητας ή για μια ε, μεταφορά σε έναν άλλο τρόπο μετατόπισαν ε, έναν άλλο τρόπο μεταφράσης. Το θέμα είναι ότι η περιβαλλοντική διάσταση δεν είναι απαραίτητο να είναι η πρωταρχική παράμετρος. Περνάμε λοιπόν ε, στα συμπεράσματα. Ποιες είναι οι σημαντικότερες τρεις οικολογικές καινοτομίες που εντοπίσαμε. Πρώτα απ' όλα, οι περιορισμοί στις εκπομπές του του άνθρακα για τα οδικά οχήματα. Δεν είναι να μιλάμε μόνο για τα αυτοκίνητα, αλλά και τα φορτηγά περιλαμβάνονται σε αυτή τη διάταξη, ε, καθώς και, τα... και οι μηχανές. Προσπαθούμε να δούμε πώς ε, τα νέα οχήματα τα οποία αγοράζονται θα μπορούσαν ε, να περιορίσουν τις εκπομπές ε, καυσαερίων. Νομίζω ότι αυτή άλλωστε είναι και η σωστή προσέγγιση που υιοθετεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση ό,τι αφορά την αγορά αυτοκινήτων. Έπειτα, δεύτερο στοιχείο, η εσωτερήκευση των εξωτερικών δαπανών, των εξωτερικών μεταφορικών δαπανών. Η χρήση των μεταφορικών υπηρεσιών οδηγεί ε, αυτοί παίρνουν, ε, επομίζονται και το οικονομικό αλλά και το περιβαλλοντικό κόστος, ε, το κόστος συμφόρησης και τα λοιπά. Άρα όλα αυτά συνεπάγονται την εσωτερήκευση του εξωτερικού κόστους και όλοι γνωρίζουμε ότι είναι μια πολιτική αυτή η οποία έχει ξεκινήσει και προωθείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα εδώ και δύο-τρεις τουλάχιστον δεκαετίες. Δεν έχει πλήρως εφαρμοστεί εξού και περιλαμβάνεται ακόμη στον κατάλογο με τα βασικά ε, σημεία μας. Και ίσως η σημαντικότερη οικολογική καινοτομία είναι η εισαγωγή ουδέτερων ως προς τον άνθρακα καυσίμων. Ορίζουμε λοιπόν και εντοπίζουμε κάποια συγκεκριμένα καύσιμα τα οποία για κάποιους τρόπους μεταφοράς θα μπορούσαν να είναι σημαντικά θα πρέπει λοιπόν η κινητικότητα να εφαρμοστεί κυρίως ε, στις οδικές μεταφορές ε, και θα αφορά τα φορτηγάκια και τα αυτοκίνητα οχήματα και θα αφορά και διάφορα μορφές, ε, τα ευρεδικά, τα ηλεκτρικά οχήματα. Αλλά από την άλλη πλευρά σε ό,τι αφορά τη χρήση των βιοκαυσίμων, νομίζουμε ότι αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται περισσότερο στις αεροπορικές μεταφορές. Τι άλλο πρέπει να αναφέρουμε για αυτές τις τρεις οικολογικέ καινοτομίες. Είναι αλληλοσυμπληρούμενες. Δηλαδή, εάν τις εφαρμόσετε ταυτόχρονα, αλληλοενισχύονται τα ωφέλη τους. Άρα, ε, έχουν ε, εκθετικό αποτέλεσμα και όχι απλά ε, και σωρευτικό. Και βέβαια θα βελτιωθεί και η προστασία του περιβάλλοντος και στο τοπικό και αστικό επίπεδο, αλλά και ο παγκόσμιος αντίκτυπος στο περιβάλλον θα είναι μικρότερος. Κάτι πολύ σημαντικό λοιπόν πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Δεύτερη ομάδα τώρα σημαντικών οικολογικών καινοτομίων. Δύο αστικές όπως τις αποκαλούμε είναι η ελπίδα μας για το μέλλον, γιατί είναι κάτι καινούριο. Πρώτα απ' όλα επιβατηγές, ε, μεταφορές επιβατών, τρόπος ή σύστημα μεταφορών που είναι εναλλακτικό και νέο στις ε, αστικές περιοχές. Δηλαδή, ο χρήστη των μεταφορών, των συγκοινωνιών μπορεί να αγοράσει τι ε, υπηρεσίε κινητικότητα, δημόσιε συγκοινωνίε ε, ή ε, κοινό αυτοκίνητο, κοινό όχημα από τον ίδιο πάροχο, ίσω και μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, για παράδειγμα. Ή μπορεί να αναπτύξει ένα επιχειρηματικά μοντέλα, την μοναπευθυντική θηρίδα. Ένας λοιπόν πάροχος κινητικότητας για τον πελάτη ο οποίος συνδυάζει διάφορους ε, παρόχους μεν, αλλά ο πελάτης έχει τη σύμβασή του με έναν μόνο πάροχο κινητικότητας. Και ένα τρίτο στοιχείο το οποίο ήδη προανέφερα είναι η συμπερίληψη, συμπερίληψη νέων ε, τρόπων. Παραδείγματο χάρη η χρησιμοποίηση ενός κοινού οχήματος και όχι η ιδιοκτησία οχήματος, το sharing και όχι το owning. Έχουμε έναν αστικοποιημένο κόσμο, όλο και περισσότερο. Θέλουμε να βελτιώσουμε την ε, ποιότητα της ζωής, ε, να είναι πιο πράσινες οι πόλεις, ε, να είναι πιο κατάλληλες, ώστε ο κόσμος να περπατάει, να χρησιμοποιεί το ποδήλατο και όχι να παίρνει το αυτοκίνητο. Είναι η λεγόμενη αντίληψη για τον πέμπτο τρόπο μεταφοράς. Εν συνεχεία, εντοπίσαμε τρεις οικολογικές καινοτομίες στον τομέα των επαγματικών μεταφορών. Η πρώτη καινοτομία σχετίζεται με την εκπαίδευση των οδηγών, φορτηγών, αλλά και των σειρμών, των ε, σιδηροδρόμων. Έχει αλλάξει το timing των μεταφορών, άρα θα πρέπει να προσαρμοστούν ε, και τα συστήματα ελέγχου. Θα πρέπει λοιπόν να προσαρμοστούν ε, στις ανάγκες της οικολογικής οδήγησης. Επίσης, θέλουμε να υπάρχουν συνεργατικές ε, μέθοδοι εφοδιαστικής logistics μεταξύ των μεταφορέων. Να υπάρχει μια δεσμοποίηση των ροών των μεταφορών, ώστε οι μεταφορές των εμπορευμάτων να είναι πιο αποδοτικοί, είτε με, καλύτερο, με πιο αποδοτικό τρόπο μεταφοράς ή με μεγαλύτερα οχήματα ή με την μεταφορά ε, στο σιδηρόδρομο ή στη ναυσιπλοεία ε, αλλά το σημαντικότερο στοιχείο το οποίο πρέπει να αναφέρουμε εδώ είναι αυτή η συνεργατική προσέγγιση, ότι θα πρέπει δηλαδή διαφορετικές εταιρείε να συνεργάζονται μεταξύ τους για να το πετύχουν αυτό. Τρίτο στοιχείο που εντάσσεται και στα άλλα δύο είναι η τριτροπική εμπορευματική διατροπικότητα. Trimodal freight intermodality. Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε τριτροπικούς κόμβους οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις επίσης θα πρέπει να μπορούν αυτές τις αντιλήψεις, αυτές τις έννοιες να τις αξιοποιήσουν. Άρα πρέπει να ενημερωθούν καλύτερα για όλες αυτές ε, τις νέες ε, ιδέες για να μπορέσουν αυτούς τους τροπικούς κόμβους να τους χρησιμοποιήσουν και να σχεδιάσουν ανάλογα και, τις, ε, και τα logistics τους. Ποια είναι η διαφορά σχέση με την πρώτη ομάδα, ότι η ίδια η βιομηχανία θα πρέπει να αλλάξει τις δομές logistics και να αυξήσει τη συνεργασία. Και η κυβέρνηση θα πρέπει να θεσπίσει τα πλαίσια για τις νέες αυτές μορφές συνεργασίας. Τέλος, δύο τελευταίες οικολογικές καινοτομίες που εντοπίσαμε και συμπεριλάβουμε στον κατάλογο των δέκα σημαντικότερων καινοτομιών είναι η σιδηρόδρομοι υψηλής ταχύτητας, η σπονδυλική στήλη λοιπόν τρένων υψηλής ε, ταχύτητας ε, και κόμβων σχετικών. Αυτό όμως δεν θα πρέπει να είναι απομονωμένο, θα πρέπει να διασυνδέεται και με την περιφερειακή πρόσβαση. Ίσως και με άλλους τρόπους μεταφοράς. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί βελτιώνει ε, την εναλλακτική μεταφορά επιβατών με άλλους τρόπους μεταφοράς. Επίσης, ε, συζητήθηκε και πριν εδώ ε, το θέμα των καθαρών ε, θαλάσσιων μεταφορών. Πρόκειται για μια δέσμη μέτρων που έχουμε περιλάβει και στη δική μας μελέτη, τεχνολογικά μέτρα, αναδιαμόρφωση τη πρόθεσης και άλλων συστημάτων των πλοίων, καθορισμός προτύπων, το Energy Design Index για παράδειγμα, που ορίζει κάποια όρια για τα πλοία τα οποία θα αναπηγηθούν στο μέλλον και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τα στοιχεία για τις καθαρές ε, θαλάσσιες μεταφορές θα βελτιώσουν και τον μείζωνα διεθνή πορευματικό τρόπο μεταφορών. Αυτά λοιπόν ε, και εδώ κάποια highlights από την online έρευνα την οποία κάναμε. είχε διάρκεια τριών-τεσσάρων εβδομάδων και ένα από τα ερωτήματα τα οποία θέσαμε στους απαντώντες ήταν ποια πιστεύουν ότι είναι τα σημαντικότερα μέτρα. Τους προτείναμε 10 μέτρα, τα σημαντικότερα σε ό,τι αφορά τη βιώσιμη κινητικότητα και ο κάθε απαντών μπορούσε να διαλέξει τρία μέτρα. Και τους δίσαμε και να τα κατατάξει σε σειρά προτεραιότητα. Πρώτο, σημαντικότερο, δεύτερο, τρίτο. Βλέπετε λοιπόν ε, την ομαδοποίηση, βλέπετε την συνολική κατάταξη τρεις βαθμούς έπαιρνε το σημαντικότερο, το πρώτο σημαντικότερο και έναν βαθμό το, εν, το τρίτο σημαντικότερο μέτρο. Και βλέπετε και τα αποτελέσματα. Σε ό,τι αφορά τώρα τα πρότυπα για τις εκπομπές της διοξιδίου του άνθρακα, αυτά θεώρησαν οι απαντώντες ως το σημαντικότερο μέτρο, ως καινοτομία και για την κινητικότητα, τη βιώσιμη. Και το δεύτερο σημαντικότερο ήταν ε, τα ουδέτερος προς τον άνθρακα καύσιμα. Δεύτερο ερώτημα, πώς οι διάφορες αυτές οικολογικές καινοτομίες μπορούν να ε, συνεργάζονται μεταξύ τους, δηλαδή είναι συμβατές μεταξύ τους ε, ή μήπως ε, αντικρουόμενες. Αναφέραμε τρεις τουλάχιστον συνεργατικές αλληλεπιδράσεις ανά μέτρο. Ποιο ήταν το πιο θετικό μέτρο ήταν η εσωτερήκευση. Και τώρα Έρχομαι σε κάποια πιο θεωρητικά στοιχεία στο πλαίσιο του αναλυτικού πλαισίου. Τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως δείκτες για την οικονομικό αντίκτυπο. Πρώτα απ' όλα η προοπτική του χρήστη. Αλλαγή του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας, διασύνδεση αυτού του κόστους ιδιοκτησίας με τις μειώσεις των θερμοκηπιακών αερίων Μπορούμε να υπολογίσουμε ένα κόστος μείωσης των εκπομπών, για παράδειγμα συχνά χρησιμοποιείται για τις οικονομικές ε, εκτιμήσεις. Επίσης, η μεσοοικονομική προοπτική, πώς αντιδρούν οι τομείς, ε, ποιες είναι οι αλλαγές στις επενδύσεις. Αυτά είναι σημαντικά θέματα και ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Χρειάζονται περισσότερες επενδύσεις ή μπορούμε να μειώσουμε τις επενδύσεις, να τις μετακυλήσουμε τις επενδύσεις κάπου αλλού. Και στην πολιτική συζήτηση, στον πολιτικό διάλογο επίσης, κάτι πάρα πολύ σημαντικό εδώ είναι και η μακροοικονομική προοπτική, ιδίω ε, στη σημερινή εποχή. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την και να τονώσουμε την ανάπτυξη και την απασχόληση. Επίση, η προοπτική τη πρόνοια, ανάλυση κόστου ωφέλου, ένα δείκτη πολύ σημαντικό και συχνά χρησιμοποιούμενο. Ε, βλέπουμε ποιε εξοικονομήσει ε, χρόνου υπάρχουν ε, με την εισαγωγή κάποιων μέτρων κτλ. Επίση, η προοπτική που αφορά τη διανομή, δηλαδή ποιοι ε, ωφελούνται, ποιες ομάδες, ε, ποια επίπεδα, περιφερειακά κτλ. Και μια νέα ε, προοπτική σημαντική για όλα αυτά τα μέτρα όμως, που βελτιώνουν, τα μέτρα αυτά που βελτιώνουν την αποδοτικότητα και την ενεργειακή κατανάλωση μπορούν να οδηγήσουν σε αλλαγή των εσόδων των κρατικών Άρα είναι και η κρατική πτυχή, η κυβερνητική πτυχή. Κάποια παραδείγματα σε ό,τι αφορά το κόστος ε, για το χρήστη. Για τα μέτρα αυτά με βάση το κόστος του, για το χρήστη είχαμε τελείως διαφορετικά αποτελέσματα. Βλέπετε, για τα πρότυπα για τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα έχουμε κέρδος 100 ευρώ ανατόνο διοξιδίου του άνθρακα. Σε ό,τι αφορά τώρα τις καθαρές θαλάσσιες μεταφορές είναι μια διαφορετική εικόνα αυτή που βλέπουμε. Με το κόστος μείωση των εκπομπών βλέπουμε από το 1.360 ε, άλλες φορές δηλαδή να έχουμε ε, απώλεια και άλλες φορές να έχουμε κέρδος, 40 παραδείγματος χάρη ευρώ. Τα βιοκαύσιμα πάντα έχουν ένα κόστος μέσα των εκπομπών, τουλάχιστον μέχρι το 2020. Ένα άλλο θέμα, σημαντικό και αυτό, στο πλαίσιο της ε, online αυτής έρευνας, Ζητήσαμε από τους ερωτώμενους να μας πούν ποιος είναι ο μακροοικονομικός αντίκτυπος των 10 μεγαλύτερων οικολογικών καινοτομιών. Τις είδαν αρκετά θετικές, τα 9 συγκεκριμένα μέτρα, τα είδαν θετικά, αλλά μόνο για την εσωτερική και του εξωτερικού κόστος. Ο μακροοικονομικός αντίκτυπος ε, εκτίμησαν ότι θα είναι αρνητικός. Εν συντομία, σε ό,τι αφορά του περιορισμού που έχουμε εντοπίσει για τι οικονομικέ εκτιμήσει, πρώτα απ' όλα ε, το επίκεντρο είναι το κόστο για το χρήστη. Η πολιτική εστιάζει επίσης ε, στις εξοικονομήσεις ε, ε, ως προς το χρόνο. Και επίσης ποιες είναι οι δομικές αλλαγές που μπορούν να γίνουν. Αυτές μακροπρόθεσμα φαίνεται ότι παραγνωρίζονται στις εκτιμήσεις. Και έρχομαι στο τελευταίο τμήμα της παρουσίασης που είναι οι συστάσεις. Έχουμε λοιπόν ομαδοποιήσει τις συστάσεις μας σε κάποιους τομείς. Πρώτα απ' όλα τεχνολογία και φόροι πρώτη ομάδα. Εδώ τι συνιστούμε λοιπόν. Φιλόδοξα όρια εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα για τα οδικά οχήματα. Αναφέρουμε εδώ συγκεκριμένα φορτηγά, και ε, αυτοκίνητα. Και έχουμε και ένα προφίλ χρονικό ώστε να μπορεί η βιομηχανία να εφαρμόσει τις αποφάσεις οι οποίες πρέπει να είναι και καλά τεκμηριωμένες και βάσιμες. Δεύτερο στοιχείο, πρέπει να εισαχθούν ε, στις οδικές μεταφορές ε, τα ουδέτερα προς τον άνθρακα καύσιμα και είπατε εδώ υπάρχει διασύνδεση και με ειδικά καύσιμα ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς. Η κινητικότητα αφορά κυρίως το e-mobility, αφορά κυρίως τις οδικές μεταφορές. Η έρευνα και η ανάπτυξη πρέπει να ενισχυθεί και για τα βιοκαύσιμα πρέπει να στηριχθούν περισσότερο για να ανοιχθούν και να εφαρμοστούν. Μιλήσαμε επίση και για τι ποσοστώσει που και αυτέ θα πρέπει να είναι δυναμικέ ώστε ρεαλιστικά να μπορούν να αυξηθούν συν το χρόνο. Και κάτι άλλο που πρέπει να έχουμε υπόψη μα είναι ότι θα πρέπει οι πολιτικές αυτές να στηριχθούν από την εσωτερική και του εξωτερικού κόστου των ορυκτών καυσίμων. Αυξάνεται το κόστος και οι φόροι αυξάνονται συν το χρόνο και οι υπόλοιπε πολιτικές θα πρέπει να προσφέρουν σε το χρόνο ελκυστικές λύσεις και κόστος μείωση των εκπομπών. Βέβαια είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στο μέλλον ε, αναμένεται και αύξηση των τιμών πετρελαίου. Δεύτερη πτυχή στο πλαίσιο των τριών αυτών μέτρων και τη εφαρμογή του είναι το χρονοδιάγραμμα, το timing. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να βαδίζουν παραλίλω. Να βελτιωθούν επίσης τα φορολογικά επίπεδα ταυτόχρονα. Και έρχομαι στην επόμενη διαφάνεια, πάντα σε σχέση με την τεχνολογία και τους φόρους. Ήδη σα ανέφερα. Αν θέλουμε να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα του τομέα των μεταφορών, και αν δούμε και τα κρατικά έσοδα από την φορολόγηση των καυσίμων, τις μεταφορές, αυτά τα έσοδα ε, θα μειωθούν δραστικά. Άρα, μια πτυχή εδώ είναι να αντισταθμίσουμε ε, αυτές ε, τις απώλειες. Είτε να αυξηθούν οι φόροι των καυσίμων ή βαθμιαία να υπάρξουν χρεώσεις για τις οδικές μεταφορές Κάνουμε κάποιες μελέτες αυτή τη στιγμή, ε, βλέποντας τις βελτιώσεις ό,τι αφορά την αποδοτικότητα στις οδικές μεταφορές. Βλέπουμε ότι υπάρχει ε, σημαντική μετατόπιση στις οδικές μεταφορές, αν δεν υπάρξει κάποια αντιστάθμιση. Εκεί βλέπουμε να μειώνεται. Δεν έχουμε τις ίδιες βελτιώσεις ε, στην αποδοτικότητα στις θαλάσσιες και στις μεταφορές. Και πέμπτος ε, τρόπος μεταφοράς είναι το επόμενο ε, slide μου και οι σχετικές ε, συστάσεις. Για να χρησιμοποιηθεί αυτός ο πέμπτος τρόπος στις διαφορετικές πόλεις της Ευρώπης το να είμαι εγώ υπάλληλο ενό παρόχου κινητικότητα ε, ε, στο Βερολίνο, αλλά να μην μπορώ να χρησιμοποιήσω τι υπηρεσίε ε, στι Βρυξέλλε ή οπουδήποτε αλλού, δεν έχει κανένα νόημα. Άρα θα πρέπει αυτό ο πέμπτο τρόπο να μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή πόλη. Θα μπορούσε να είναι ένα είδο ε, περιαγωγή στον τομέα τη κινητικότητα και των μεταφορών. Αναφέρουμε επίσης παράλληλα ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής της πόλης και παρατηρήσαμε ότι με κάποια μέτρα πράγματι συμβαίνει αυτό. Ένα από αυτά τα ε, προγράμματα που μπορούν να εφαρμοστούν είναι τα βιώσιμα αστικά σχέδια κινητικότητας και τα σχέδια μείωσης ε, της ηχορύπανσης. Κυρίες, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να συνεχίσω ε, είμαι ο Βέρνερ ε, Ρότεν Γκάτερ από το KIT, από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καρτσρούης. Ε, Θα ασχοληθώ με το δεύτερο τμήμα της ε, μελέτης που αποδεικνύει ότι ε, υπάρχει υποτίμηση ε, της μείωσης των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος και άλλων οχλήσεων σε σχέση με την επίπτωση που θα είχαν στην ποιότητα ζωής γενικότερα. Υπάρχουν, πρέπει να υπάρχουν προγράμματα εκπαίδευσης. Πώς εκπαιδεύεται κανείς για να μάθει να οδηγεί ή στις ε, εσωτερικές πλωτές οδούς ή στους σιδηροδρόμους. Και το δεύτερο είναι η κοινή επιμελητία, δηλαδή ε, να οργανώνουν τα logistics την επιμελητία κάποιες εταιρείε από κοινού. Με τον τρόπο αυτό γίνεται εξοικονόμηση ενέργειας ε, και περιβαλλοντικής μόλυνσης. Τρίτο στοιχείο είναι η ενδυνάμωση των διατροπικών κόμβων, intermodal hubs. Βεβαίως το βέλτιστο είναι να έχει κανείς και τα τρία αυτά στοιχεία έτσι ώστε να μειωθεί σημαντικά ε, η εκπομπή διοξιδίου του άνθρακος αλλά και της περιβαλλοντικής μόλυσης γενικότερα. Πιστεύουμε ότι ε, έχει παραμεληθεί το θέμα αυτό τον τελευταίο καιρό, γιατί πρώτον ε, έχουμε πάρα πολύ γρήγορη ανάπτυξη και επομένως ε, ε, κάθε μέτρο το οποίο αποσκοπεί στην ε, πρασινότερη ας πούμε μεταφορά ε, ξεπερνιέται από την ίδια την ανάπτυξη που είναι διπλή σε σχέση με το ΑΕΠ το ε, ΑΕΠ μπορεί να αυξηθεί κατά 1,5% ενώ ας πούμε οι μεταφορές το ΦΡΕΤ ε, κατά 3%. Επομένως καταλαβαίνετε ότι ε, πολύ γρήγορα προχωρούν οι μεταφορές έστω και αν στο μέλλον υπάρχει πρόβληση επιβράδυνσης της ανάπτυξης του ΑΕΠ πολλοί εμπειρογνώμονες ε, πιστεύουν ότι τα μέτρα μετριασμού ε, μπορεί να έχουν ε, λιγότερη επίπτωση στην μεταφορά και γι' αυτό λοιπόν αυτού του είδους τα μέτρα δεν αναφέρονται πολύ συχνά στην μεταφορά εμπορευμάτων. Δεν παίζουν, η μεταφορά εμπορευμάτων δεν παίζει πολύ σημαντικό ρόλο Επίσης, τα, υπάρχουν αποθέματα τα οποία παραμένουν ανεκμετάλλευτα ε, ε, όσον αφορά την οργάνωση. Και επομένως ε, σας έδωσα ένα παράδειγμα αυτήν την κοινή, τη μοιρασμένη επιμελητία και αναφέρω και άλλα στοιχεία βεβαίως στην μελέτη μας. Πάντως η από κοινού επιμελητία μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους, δηλαδή ε, να γίνουν ε, όμιλοι επιχειρήσεων. Ε, δεύτερον, μπορεί κάποιες μικρές ή μικρομεσαίες επιχειρήσεις να επιλέξουν τον ίδιο πάροχο υπηρεσίας, δηλαδή έναν ανεξάρτητο πάροχο επιμελητίας ε, και όλοι να ε, από να αποτανθούν σε αυτόν τον πάροχο. Και υπάρχει ένας τρίτος τρόπος οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να έχουν κοινή επιμελητία με τους προμηδευτές. Και ε, καταλαβαίνετε ότι με τον τρόπο αυτό ε, μπορούν να μειωθούν ε, οι τιμές. Το 2006 ε, έγιναν κάποιες πρώτες προσπάθειες ε, οι εταιρείε μαζί με τους πάροχους να έχουν κοινή επιμελητία και πραγματικά έδωσε τα καλύτερα αποτελέσματα. Ε, οι εταιρείε κέρδισαν χρήματα και χρόνο και η κοινωνία κέρδισε λιγότερη μόλυνση. Αυτά είναι κάποια ε, σημεία εκκίνησης. Μπορεί κανείς όμως να βρει πάρα πολλά παρόμοια στοιχεία. Ε, η, ε, αυτή η κοινή επιμελητία είναι μια προσπάθεια προσωπικής βελτίωσης υπάρχουν και άλλες ε, ε, δυνατότητες ομαδοποίησης ε, επιχειρήσεων και επιχειρηματικών διαδικασιών. Οι ίδιες οι εταιρείες μπορούν να βρουν τον τρόπο με τον οποίο να αναπτύξουν κοινά προγράμματα στο μέλλον. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε ότι τα επιτεύγματα και όσον αφορά ε, στην μεταφορά εμπορευμάτων και σε ε, άλλα ε, αναφέρονται σε πολλά εργαλεία. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν, είναι πολύ καλύτερα να χρησιμοποιηθούν και τα δέκα εργαλεία μαζί έτσι ώστε να έχει κανείς την, δυνατότη, την καλύτερη δυνατή απόδοση. Απ' την άλλη πλευρά, ε, εάν ας πούμε μιλάμε για αύξηση των φόρων Προφανώς δεν είναι δυνατόν ε, μόνο με αυτό το μέτρο να εξηγιανθεί η κατάσταση. Δεν είναι δυνατόν όλες οι ασθένειες να έχουν μόνο μία θεραπεία και αυτό να είναι ε, η φορολόγηση. Ίσως να είναι ο απλούστερος ε, τρόπος, αλλά παρόλα αυτά δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δηλαδή θα πρέπει ταυτοχρόνως με την φορολόγηση να υπάρχουν και, άλλες, και άλλα μέτρα η τι σημαίνει πολιτική και τα Οδηγούμε λοιπόν στο επόμενο σημείο μου που είναι οι μελλοντικέ προκλήσεις. Δεν είναι δυνατόν να ανταποκριθούμε ε, στο, στα ανάγκες του και τις απαιτήσει του μέλλοντος ε, εάν δεν προσαρμοστούμε. Αναφέρθηκα προηγουμένως ε, στην δημιουργία σημαντικών διατροπικών κόμβων χρειαζόμαστε ε, μεγαλύτερη ομαδοποίηση, χρειαζόμαστε ε, επομένως ένα καλύτερο ε, δίκτυο κόμβων που θα έχουν και άμεσο και έμεσο αντίκτυπο. Δηλαδή θα υπάρχει οπωσδήποτε μείωση κόστους, θα υπάρχει οπωσδήποτε μείωση χρόνου κέρδος επομένως και στις δύο περιπτώσεις, άρα καλύτερος λόγος κέρδους κόστους ε, ωφελίας ε, και ε, βεβαίως αύξηση της ανταγωνιστικότητας και φυσικά καλύτερη ασφάλεια ενεργειακή όσο και οι πόροι γίνονται όλο και πιο σπάνιοι. Αυτό σημαίνει, και εδώ έρχομαι στην αξιολόγηση, αξιολόγηση με προγραμμάτων όπως ε, είναι τα ε, δίκτυα TNT. Ο μακροχρόνιος στόχος θα πρέπει να είναι το πρώτο μέλημα και όχι τόσο τα ε, βράχη πρόθεσμα ωφέλη για τους χρήστες. Αυτή η ολιστική αντιμετώπιση είναι τελικά πιο επωφελής για τους χρήστες. Επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η επιχειρηματικότητα θέλει και οι επενδύσεις θέλουν διαρκή ε, ερεθίσματα. Επομένως και εδώ θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε ε, αποτελεσματικότερα τις μακροχρόνιες τροποποιήσεις ε, του, της μορφής ε, των ε, μεταφορών. Γιατί το πρόβλημα παραμένει πάντα το ίδιο. ε, ε με τις στατιστικές του παρελθόντος βλέπεις το παρελθόν, ενώ πρέπει κανείς να κάνει προβολή για τα επόμενα 20-30 χρόνια, πάντα προβολή στο μέλλον. Ε, ε, πολλές φορές ε, οι οικονομικές αποτυχίες προέρχονται βεβαίως από λανθασμένες εκτιμήσεις αλλά και από την αστάθεια. Χρειάζεται λοιπόν ένα περιβάλλον σταθερότητας, ένα περιβάλλον βεβαιότητας και για να γίνει αυτό πρέπει κανείς να έχει σαφή εικόνα για το μέλλον, ένα σαφές ε, ε, σχέδιο ε, για το μέλλον και βεβαίως εδώ να ενταχθούν και τα προβλήματα, οι φορείες τα οποία αναφέρθηκαν και προηγουμένως. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω βεβαίως για την προσοχή σας, αλλά ε, παρόλα αυτά ε, θα ήθελα να πω ότι ε, οι επενδύσεις σε καλύτερο περιβάλλον στον τομέα των μεταφορών όχι δεν οδηγούν μονάχα σε καλύτερες μεταφορές αλλά οδηγούν και σε νέες διαδικασίες, σε νέες αγορές, σε νέα προϊόντα. Είναι επομένως απαραίτητη για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας στην παγκόσμια αγορά. Επομένως, εάν θέλουμε να είμαστε μέρος των, ε, ε, των διεθνών συναλλαγών θα πρέπει να κάνουμε κάποια βήματα διορθωτικά. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Ευχαριστώ πολύ τους δύο μιλητές, τον κύριο και τον κύριο Ρόπιν Κάτσα. Προσπαθώ να συμβαστώ με την ιδέα ότι δεν πρόκειται να τελειώσουμε νωρίς όπως ήθελα. Γιατί όλα και περισσότερο το λόγο. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν. Ο κύριος Γκρός έχει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο μιλητές για την παρουσίαση των θεμάτων. Μένουν θέματα σημαντικά να συζητήσουμε τις, ενέργεια, τις ε, ουδέτερες ως προς το διοξείδιο του άνθρακα ενέργειες που χρειαζόμαστε. Και βέβαια το θέμα αυτό σε συνδυασμό με τις εσωτερικές μετακινήσεις. Μίλησατε επίσης για συνεργασία μεταξύ μικρότερων και μεγαλύτερων επιχειρήσεων καλύτερο συντονισμό των μεταφορών. Αν κατάλαβα καλά, θεωρείτε ότι και, και τα πράσινα λεωφορεία μπορεί να είναι χρήσιμα ή κατάλαβα λάθος ενδεχομένω. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε εν γέννη με το θέμα της ε, ανάπτυξης της συνδυασμένης με την κινητικότητα και τις μεταφορές. ένα καλό επιχείρημα, ένα οικονομικό επιχείρημα. Και γι' αυτό θα ήθελα να μου πείτε ποιες είναι κατά την άποψη σας οι πιο καλές προσεγγίσεις για να μπορέσουμε να προαγάγουμε αυτά τα μιλήματα. Ο κύριος Ολκαντράουι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ τους δύο μίλητες. Προφανώς μόλις έλαβα και εγώ την έκθεση στα χέρια μου αν κατάλαβα καλά όμως είναι μάλλον προσωρινή αυτή η έκδοση. Προσωρινή η οποία είναι μονιμότερη της θελικής. Γι' αυτό λοιπόν ερωτώ εάν σκοπεύετε να κάνετε κάποιες σοβαρές τροποποιήσεις ή αν είναι πράγματι το οριστικό κείμενο λίγο πολύ αυτό που θα δούμε. Και γέννη θα ήθελα να πω ότι ε, ιδιαίτερα εκτιμώ τα όσα μας είπατε στις προτάσεις σας. Έχετε καταγράψει μια σειρά δηλαδή από πράγματα, δυνατότητες ε, που προσφέρονται για να, για να καταστήσουμε τις μεταφορές μας πιο βιώσιμες. Είπατε και εσείς ε, διάφορες προτάσεις, αναφέρατε διάφορες προτάσεις, οι οποίες όντως μας απασχολούν και εμάς εδώ στο Κοινοβούλιο. Ερωτώ λοιπόν εάν υπάρχει πρόθεση για την ε, μεταφορά επιβατών, αυτό που αναφέρατε ως πέμπτο μέσο, πέμπτο τρόπο μεταφορών, και επίσης προτάσεις σας για τις ε, μεταφορές. Βλέπω αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα, δυστυχώς όμως δεν έχει προχωρήσει αρκετά η εξέλιξη. Για τη μεταφορά των εμπορευμάτων ωστόσο και στα όσα είπε και ο κύριος ε, Γκρός. Μιλάτε για συνεργασία, λέτε ότι μπορούμε από τη συνεργασία αυτή να αποκομίσουμε αρκετά ωφέλη. Ερωτώ λοιπόν πώς μπορεί να γίνει πιο ελκυστική η συνεργασία σε τι δράση μπορούν να αποδυθούν ε, οι δημόσιες αρχές, τι χρειάζεται να πράξουν οι δημόσιες αρχές, ε, Φερπίν με την επιβολή υψηλότερων τιμών ε, μπορούμε να ζητήσουμε, μπορούμε να περιμένουμε καλύτερη συνεργασία, να υποχρεωθούν δηλαδή λόγω των τιμών οι εταίροι να συνεργαστούν περισσότερο. Η κυρία Σουνέρ, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση. Θα ήθελα να φέρω τέσσερις συγκεκριμένε ερωτήσεις, ε, παρατηρήσεις. κάτι που δεν έχω καταλάβει στο Ε, κείμενό σας το σχετικό με το κόστος του ε, διοξιδίου του άνθρακα ανατόνο όπου λέτε ότι στις θαλάσσιες μεταφορές υπάρχει ε, θέμα κόστους 62-4 ευρώ ανατόνο διοξιδίου του άνθρακα. Τι σημαίνει ακριβώς αυτό. Μετά, θα ήθελα να ρωτήσω αν μιλάτε μόνο για μεταφορές αστικές λεωφορεία και το καθεξής ή εννοείται και άλλα μέσα μεταφορών, ποδήλατα ή και συμπληρώνω ενδεχομένως ηλεκτρικά μέσα μεταφορών. Η αναφορά επίσης στα τρένα υψηλής ταχύτητας δεν θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνει και τα περιφερειακά τρένα της περιφερειακής συνδρομικές συνδέσεις. Η ανάπτυξη της υπαίθρου πρέπει να προσβα λάβει περισσότερη σημασία στην έκθεση σας πιστεύω, διότι ε, η χωροταξία θα πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ε, ρόλο εδώ πέρα, η ανάπτυξη της υπαίθρου για η χωροταξία. Και επίσης οικονομικά και οικολογικά συστήματα ευφυή μπορούν να βοηθήσουν στην αποφυγή των κυκλοφοριακών συμφορήσεων, στην αποσυμφέρηση των δρόμων και όλα αυτά. Αλλά έχετε κάτι συγκεκριμένο να προτείνετε. Μιλάτε για καινοτομία, αλλά όχι σε αρκετέ λεπτομέρειε. Κύριο Κράμερ. Φυσικά ευχαριστώ και εγώ τους δύο μελητές για τη μελέτη τους, για την παρουσίαση. Είναι πολύ χρήσιμη. Η έννοια του immobility, της ακινησίας δηλαδή, δεν είναι καινούρια. Την, ε, το φαινόμενο αυτό το παρατηρείται ήδη το 1980 στο Βερολίνο. Και πιστεύω ότι θα πρέπει και για την ε, κινητικότητα μέσα στις, ε, στα αστικά κέντρα να ζητήσουμε λύσεις πιο πρωτότυπες, γιατί ακόμη και το ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι αθώο, έχει εξίσου επιβαρυντική δράση όσο και άλλα μέσα μεταφορών στην αλυσίδα του. Θα ήθελα λοιπόν επίσης μια και διαφοροποιείται μεταξύ βράχη και πρόθεσης προσέγγισης, να επισημάνω ότι από τη συνδρομική μεταρρύθμιση στις, στη Γερμανία έχουμε επενδύσει 40 δισεκατομμύρια στις ε, μεγάλων αποστάσεων ε, μεταφορές, έχοντας όμως παραμελήσει σημαντικά της, ε, την Ήπεθρο. η οποία όμως η πεθρώση μετακίνηση, δηλαδή προς και από, ε, παρουσιάζει στην ε, ουσία αύξηση κατά ποσοστό έως και 50%. Μήπως λοιπόν εδώ έχουμε κάνει το λάθος του προσανατολισμού που θα έπρεπε να αλλάξουμε προσέγγιση. Το ίδιο και με τις θέσεις εργασίας. Ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες το φαινόμενο που παρατηρείται είναι πολύ μεγάλα αστικά κέντρα, στα οποία αν δεν έχει κανείς αυτοκίνητο δεν μπορεί να μετακινηθεί, δεν μπορεί να πάει στη δουλειά του καν. Ενώ μπορούμε να έχουμε εμείς μια διαφορετική προσέγγιση με μικρότερες αποστάσεις, με αποστάσεις τέτοιες που μπορεί κανείς με τα πόδια να πάει να κάνει τα ψώνια του στον μπακάλι και ως εκ τούτου να επιβαρύνει και λιγότερο το περιβάλλον, αλλά και γενικότερα την οικονομία αυτή, δηλαδή διαφορετική οικονομική προσέγγιση με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και επίση η συνεργασία. Είπατε ότι όταν άρχισαν να ανεβαίνουν τιμέ του πετρελαίου, άρχισαν οι μεγάλε επιχειρήσει να συνεργάζονται. Στην ε, Ελβετία όμω πρέπει να σα πω ότι αυτό γίνεται όχι μόνο λόγω τη αύξηση των τιμών του πετρελαίου, αλλά και διότι θεωρούν ότι δεν Υπάρχει λόγος να επιβαρύνουν το περιβάλλον τους ε, κατά τρόπο περιττό και έτσι αν μια μεγάλη εταιρεία μεταφορών θέλει ένα φορτηγό, θέλει μάλλον να στείλει ένα φορτηγό με εμπόρευμα από τη μια μεριά στην άλλη, θα τηλεφωνήσει στην άλλη εταιρεία για να ρωτήσει αν περισσεύει κανένα κυβικό χώρο στο δικό τη φορτηγό που τόσο άλλω κάνει το δρομολόγιο για να μην επιβαρυνθούν περισσότερο οι ε, μεταφορές και το περιβάλλον. Γιατί λοιπόν να μην γίνει αυτό και γιατί επισημαίνεται τη συνεργασία μόνο ως απόρρια της αύξησης των τιμών του πετρελαίου. Θα μπορούσε να γίνει ούτως ή άλλως και παρά τον ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων μια πρόταση για καλή συνεργασία μεταξύ αυτών. και επίσης ό,τι είδου ε, εξοικονόμηση εκπομπών και να επιδιώκουμε, μόνο αν εγκαταλείψουμε το αυτοκίνητο, δηλαδή πάμε με τα πόδια με το ποδήλατο, μπορούμε πραγματικά να απαλλάγουμε από αυτέ. Η κυρία Ντουιχόν. Ναι, μιλήσατε για πόλεις και νομίζω ότι πολύ καλά κάνετε, γιατί ακριβώς εκεί επικεντρώνεται ο πολύς ε, μετρήσατε την δυνατότητα μέσω ε, ουσιώδους αλλαγής του τρόπου μεταφοράς, ε, του τρόπου οργάνωσης των εμπορικών συναλλαγών και των μεταφορών μπορούν να δημιουργηθούν διαφορές, ας πούμε, ε, μπορέσαμε να δείξουμε ότι ε, υπήρξε δημιουργία θέσεων εργασίας ε, σε τομείς πολύ σημαντικούς που προέκυψαν μετά από τις μελέτες ενεργειακής αποδοτικότητας. Στην προκείμενη περίπτωση μπορούν να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Λοιπόν, Κοιτάξτε, θα σας δώσω τη δυνατότητα να απαντήσετε. Όταν, αρχίσετε, όταν με δείτε να κουνάω το σφυρί μου, θα ξέρετε ότι πρέπει να σταματήσετε. Θα προσπαθήσω να ξεκινήσω εγώ και μάλλον θα ε, δώσω τη σκητάλη μετά και στον συναδελφό μου. Σε ό,τι αφορά την τελική εκδοχή, την οριστική εκδοχή, αυτή τη θεωρούμε εμείς αρκετά οριστική. Βέβαια θα εξαρτηθεί και από τα σχόλιά σας αυτό. Αν γίνουν ε, δραστικά σχόλια, ίσως πρέπει να την ε, επανεξετάσουμε και την εκδοχή αυτή. Γι' αυτό δεν είναι ακόμη οριστική. Δεύτερο ερώτημα για τα ηλεκτρικά οχήματα. Και πάλι είναι πολύ σημαντικό να δούμε το χρονοδιάγραμμα, το timing, οι αποφάσεις για την αναδιάρθρωση των ενεργειακών συστημάτων στην Ευρώπη και συγκεκριμένα σε διάφορες χώρες είναι ξεκάθαρα. Πηγαίνουμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μεγαλύτερη αποδοτικότητα και ενεργειακή απόδοση, υψηλό μερίδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πολλές χώρες λένε για το 2020 να έχουμε 25 με 30% ΑΕΠ και ίσως το 2030 ακόμα περισσότερο, ίσως και κατά το ίμιση να είναι ΑΕΠ. Θα δούμε τι θα γίνει, ε, θα δούμε ποιο είναι το πιο αποδοτικό. Και κάτι άλλο που πρέπει να εξετάσουμε είναι ποιος είναι ο σωστός τρόπος, αν είναι με ισοσορευτεί το ηλεκτρικό όχημα όταν έχουμε 1,5 τόνο μάζα οχήματο στο πλαίσιο του ICE και ηλεκτρικό κινητήρα, ε, δεν ξέρω, ένα μικρότερο όχημα ε, για την πόλη, ίσως 500 ε, κιλά και κάποιες άλλες πρώτες ύλες και αλλάζει εικόνα τελείως μετά για τα ηλεκτρικά οχήματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις καθαρές θαλάσσιες μεταφορές, αριθμητικά στοιχεία. Για το κόστος ε, που σας ε, μίλησα, είπα ε, ότι είναι διαφορετικά τα μέτρα έξω και είναι και διαφορετικά τα νούμερα. Κάπου είναι αρνητικά και κάπου είναι θετικά. Άλλα μέτρα έχουν αυτό το κόστος της μείωσης των εκπομπών και άλλα δεν το έχουν. Έξω και βλέπουμε το, το όφελος ή τη ζημία, θέλετε. Και σε ό,τι αφορά το ITS, Ένα από τα μέτρα, ο πέμπτος τρόπος μεταφοράς, ε, τουλάχιστον, εκεί θεωρούμε ότι είναι σημαντικό το ITS. Αυτό αφορά τα κινητά επικοινωνιακά εργαλεία για τις ε, κρατήσεις, για το car sharing, για τις ηλεκτρονικές ε, ε κρατήσεις, ηλεκτρονικά εισιτήρια και στις δημόσιες συγκοινωνίες, ε, στο car sharing μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα ηλεκτρονικά εργαλεία υπηρεσίες ITS. Δεν μιλάμε για την ε, ε, καθοδήγηση, την κατεύθυνση των ροών, αλλά για τη χρήση αυτών των εργαλείων. Είναι σημαντικός ο χώρος, νομίζω, μπορεί να καταλάβει το ITS. Αυτό το οποίο δεν συζητήσαμε και έχετε δίκιο, είναι αυτά τα συστήματα για το traffic steering, για την κατεύθυνση της ε, κίνησης, της κυκλοφορίας. Να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Ρότεν Ε, λοιπόν, Πρώτα απ' όλα να επανέλθω στο ερώτημά σας σε ό,τι αφορά τα μεγαλύτερα οχήματα. Αν είναι λύση τα μεγαλύτερα οχήματα. Μακρύτερο, ε, μακρύτερα οχήματα. Το θέμα είναι τι είναι πιο παραγωγικό για τις οδικές μεταφορές. Με τα τεράστια φορτηγά αυτά, τα giga liners, θα αυξηθεί ε, η παραγωγικότητα κατά 25% και μπορεί να μειωθεί όμως το καύσιμο ανά τόνο κατά 15 20%. Αλλά υπάρχουν και άλλες ε, παρενέργειες, τις οποίες δεν έχουμε καταγράψει και απαριθμίσει, αλλά μπορούμε να τις συζητήσουμε και εδώ στο Κοινοβούλιο, αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Η λύση μας λοιπόν δεν ήταν να ζητήσουμε να χρησιμοποιούνται αυτά τα giga liners, αυτά τα τεράστια φορτηγά, αλλά να υπάρχει διαλειτουργικότητα μεταξύ συστημάτων και διατροπικότητα μεταξύ της εσωτερικής ε, ναυσιπλοείας, των ε, οδικών και των συνδρομικών μεταφορών. Υπάρχουν ε, κάποιες μικρές αποστολές που ομαδοποιούνται, δεσμοποιούνται και με παλέτες μεταφέρονται με τρένα στις, ε, προς προορισμούς. Έτσι έχουμε ένα συγχρονισμένο σύστημα εμπορευματικών σειρμών που έχουν όμως ίσως και καλύτερη ποιότητα, αν όχι την, τουλάχιστον την ίδια με τις οδικές μεταφορές. Αυτή είναι η λύση μας λοιπόν, η οικοδόμηση ενός ε, συστήματος ε, με συνδρομικούς κόμβους και κόμβους διασύνδεσης. Ανάλογα βέβαια με το πώς είναι και η γεωγραφία της κάθε χώρας, άλλες χώρες μπορεί να μπορούν να εκμεταλλευτούν περισσότερο τις ε, εσωτερικές πλατές οδούς, άλλες όχι τόσο. Επίσης, ε, αν έχουμε ένα συγχρονισμένο σύστημα, το οποίο συλλέγει και έπειτα ε, διανέμει και μπορούμε να έχουμε και ταυτόχρονα τα λεγόμενα main runs, δηλαδή τη βασική μεταφορά που γίνεται όλο και περισσότερο από τους σιδηροδρόμους στην προκειμένη περίπτωση. Άρα αυτή η λύση είναι η δική μας ε, ε, προτιμότερη λύση αντί για, τις, για, τη, τα μεγαλύτερα φορτηγά. Το decoupling τώρα, η απόζευξη Αν μπουν χρεώσει στι οδικέ μεταφορέ, ίσω υπάρξουν κίνητρα για την απόζεξη. Ένα ε, παράδειγμα είναι ο γαλλικό οικολογικό φόρο που σχεδιάζεται όχι για του αυτοκινητοδρόμου μόνο, αλλά 12-40.000 χιλιόμετρα του δευτερογενού ε, συστήματο. Με το σύστημα αυτό θα μπορούσε να παράσχει κανείς τα σωστά κίνητρα προς αυτήν την κατεύθυνση του decoupling ε, της αποσύνδεσης, απόζευσης. Η συνεργασία τώρα, ποιος συνεργάζεται, ποιος το κάνει, αυτό είναι ένα ερώτημα. Είτε δίνει η αγορά κάποια κίνητρα και αυτό ήταν και το επιχείρημα που ε, παρουσίασα εγώ. Η αγορά δηλαδή ανακαλύπτει πλέον αυτή την επιλογή. Το κράτος μπορεί και αυτό να βοηθήσει όμως για να επιταχυνθεί όλη η διαδικασία. Τι μπορεί να γίνει λοιπόν πρώτα απ' όλα. Να στηριχθούν τα κόνσεπτ, οι έννοιες αυτές τα rail για τα οποία σας μίλησα, αυτή η συνδρομική κόμβη, Αυτό μπορεί να το αναπτύξει μια εταιρεία, αλλά να έρθει σε σύγκρουση με το ρυθμιστή. Άρα έχουμε εδώ ένα δημόσιο στοιχείο. Ο οικοδόμηση δικτύων ενό συστήματος κόμβων έχει και μια δημόσια διάσταση, κρατική διάσταση. Άρα θα πρέπει να υπάρχει συνεκτικότητα και συνέπεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν είναι μόνο γερμανικοί σιδηρόδρομοι, παραδείγματο χάρη, που θα πρέπει να δημιουργούν αυτού του είδου το κόνσεπτ, αυτού του είδου την ιδέα. Θα πρέπει ο σχεδιασμό να γίνει εναρμονισμένα, με εναρμονισμένο τρόπο. Και χρειάζονται και περισσότερα πιλωτικά σχέδια που θα δείξουν ε, στη βιομηχανία τα πλεονεκτήματα ενό τέτοιου συστήματο. Άρα, καλό θα ήταν να ξεκινήσουν πιλωτικά κάποια προγράμματα και να μην ξεκινήσουν ε, κάποιες διαδικασίες ε, μόνο με τη χορήγηση επιδοτήσεων. Το ερώτημα του κύριου Κράμερ, μήπως έχουμε επενδύσει στο παρελθόν προς τη λάθος κατεύθυνση, δηλαδή στην κυκλοφορία μακρών αποστάσεων και όχι στις περιφερειακές τόσο συγκοινωνίες και μεταφορές και αναφέρατε και αρκετά στατιστικά στοιχεία. Δεν είναι λάθος, αλλά είναι παραπλανητικά αυτά τα στατιστικά στοιχεία. Γιατί είχαμε αυτή την αλλαγή καθεστώτος στη δεκαετία του 90, την περιφερειοποίηση των μεταφορών. Άρα μέρη των μεταφορών ε, των ε, διαστιακών Intercity έγιναν περιφερειακές μεταφορές. Μετασχηματίστηκαν σε μετα... περιφερειακές και αυτό δημιουργεί αυτή τη μεροληψία στα στοιχεία. Να μειώνονται δηλαδή οι μεταφορές μακρών αποστάσεων. Δεν συμβαίνει αυτό όμως ε, στην πράξη. Έχει αυξηθεί η συνδρομική μεταφορά μακρών αποστάσεων ιδίως ε, στις ε, νέες ε, γραμμές υψηλής ταχύτητας. Πάρα πολύ μεγάλη αύξηση παρατηρείται σε αυτό το κομμάτι των μεταφορών. Εντυπωσιακότερη μάλιστα εκεί που οι χώρες έχουν θεσπίσει πιο μακρύς διαδρόμους για τις υψηλές, για τις υψηλές μεταφορές. Άρα φυσικά και δεν ήταν άχρηστη η επένδυση στις μεταφορές και μακρών αποστάσεων και θα χρειαστεί και στο μέλλον να υπάρξει σχετική επένδυση. LSVA. Είναι ένα σύστημα χρέωσης στην Ελβετία. Αλλά αφορά πιο πολύ ε, τον τροπικό διαχωρισμό, το modal split. δεν θέλουμε να αυξηθεί η οδική κυκλοφορία. Η κυβέρνηση ε, θέλει να ακολουθήσει την πρωτοβουλία και να επενδύσει ε, στους ε, σιδηροδρόμους, στις σύραγγες, να χρηματοδοτήσει τις επενδύσεις αυτές. Και σε μεγάλο βαθμό χρηματοδοτούνται οι επιχειρήσεις από τα έσοδα. Και οι φόροι, οι χρεώσεις μάλλον, δηλαδή είναι τριπλάσιες σε σχέση με τις γερμανικές τα διόδια τα γερμανικά, που ήδη είναι αρκετά υψηλά σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Άρα νομίζω ότι είναι αδύνατον τα επόμενα χρόνια να εισαχθούν αυτά τα υψηλά ε, διόδια, υψηλέ χρεώσει που έχει εισαγάγει η Ελβετία σε όλη την Ευρώπη. Αυτό θα το δείτε και από πολιτική πλευρά είναι δύσκολο. Και βέβαια ε, πρέπει να υπάρξει και απαραίτητα αποδοχή, πάρετε πολιτική αποδοχή με την υψηλότερη τιμή λύνονται προβλήματα, αλλά δυστυχώς δεν μπορούν να υλοποιηθούν, Γιατί δεν υπάρχει μια κατάλληλη αποδοχή από την κοινή γνώμη για τα μέτρα αυτά. Ω εκ τούτου μπορούμε να σκεφτούμε το ενδεχόμενο επέκτασης αυτών των χρεώσεων, επέκτασης όχι εισαγωγής ε, των αυτοκινητοδρόμων σε ένα σύστημα χρέωσης, αλλά επέκταση, για να έχουμε δίκαιο ανταγωνισμό μεταξύ τρόπων μεταφορά. Γιατί και άλλοι τρόποι μεταφορά πρέπει να πληρώσουν για την τοπική και την περιφερειακή υποδομή. Δεν νομίζω όμω ότι μπορούμε να φτάσουμε στα ελβετικά μεγέθη των χρεώσεων. Τώρα, σε ό,τι αφορά τι νέε θέσει εργασία, ένα ερώτημα που Φυσικά, ο στόχο μα δεν είναι να καταστρέψουμε την απασχόληση, αλλά αντιθέτω να δημιουργήσουμε νέου τομεί ε, για απασχόληση έχουμε κλασικούς τομείς ανάπτυξης που ανακαλύπτει η βιομηχανία. Υγεία και περιβάλλον. Η Siemens, η General Electric για παράδειγμα, επενδύουν. Επενδύουν συγκεκριμένα σε αυτά τα ε, κομμάτια της αγοράς, γιατί θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ ψηλοί οι συντελεστές ανάπτυξης σε αυτούς τους τομείς. Και ιδίω οι συγκεκριμένοι τομείς επηρεάζονται από το κράτος σε πολύ μεγάλο βαθμό. Υπάρχει μεγάλη ευθύνη του κράτους, το οποίο θα πρέπει να ορίσει το σωστό πλαίσιο για να μπορέσουν να αυξηθούν τα θέματα αυτά της αγοράς και να αναπτυχθούν περαιτέρω. Ευχαριστώ. Ε, θα σας παρακαλούσα πολύ σύντομα. παρακολούσα πολύ σύντομα, κύριε Σόντερ. Ναι, δύο σημεία. Αναφερθήκατε στη μεταφορά void and shift. Ε, κάποια από τα μέτρα τα οποία προτείνουμε, χωρίς να μπορούμε να είμαστε βέβαια πάντα απόλυτοι και στο, στην εσωτερικοποίηση φερειπίνη σε πολυτουργικέ μεταφορέ, νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε καλές απαντήσεις και έτσι να, με, να μειωθούν ε, οι μεταφορές με το αυτοκίνητο, εφόσον προσφέρονται καλύτερες προϋποθέσεις μεταφοράς. Βέβαια αυτό θα πρέπει να ελεγχθεί κάθε φορά γιατί αν ταξιδεύουν 4-5 άτομα στο ίδιο αυτοκίνητο ή αν μεταφέρεται κάποιο φορτίο μέσα στο αυτοκίνητο ίσω να μένει αυτό πιο ε, συμφέρουσα μέθοδος μεταφοράς. Δεύτερη ερώτηση. Μας είπατε ότι δεν αναφερθήκαμε στις ε, περιοχές της Υπέθρου στο κεφάλαιο για τα τρένα υψηλής ταχύτητας. Οι εξελίξεις που περιμένουμε για την ύπεθρο στο σύστημα των μεταφορών θα είναι πολύ πιο περιορισμένες. Οι διαφορές δηλαδή σχέση με την κατάσταση θα είναι πολύ πιο περιορισμένες σε σχέση με αυτό που αναμένεται ε, σαν αλλαγή στις συνθήκες στα αναστικά κέντρα. Γι' αυτό έχουμε λιγότερη έμφαση δώσει στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ λέει ο Πρόεδρος και ευχαριστώ και τον ε, κύριο Σάντα και τον κύριο Ρότενχοφερ για την παρουσίαση αυτής της εκθέσεως σήμερα, Ρότεν Κάτσαρ, την, ε, ε, για την παρουσίαση της εκθέσεως. Ευχαριστώ τους συναδέλφους ε, επίσης για τη συμμετοχή τους. Και αν, όπως είπατε, είναι προσωρινή έκθεση, περιμένουμε στην οριστική της μορφή να συμπεριλάβετε, να ενσωματώσετε και τις ερωτήσεις και παρατηρήσεις των συναδέλφων. Ευχαριστώ πολύ, λοιπόν για, τους λοιπούς, ε, για τα λοιπά μέλη της Επιτροπής μας. Υπενθυμίζω ότι συνεχίζουμε στις 3 το απόγευμα. Με το TNT, με τα M και τον Επιτροπο Κάλλας. Πρέπει να δούμε βέβαια πώς θα το διαρθρώσουμε όλο αυτό. Σήμερα και αύριο ως προς το χρόνο μας. Θα είμαστε αυστηροί με το χρόνο λοιπόν. Γι' αυτό και θα υπενθυμίσω ότι δεν θα σας επιτρέψω να ε, μιλάτε για πάνω από πέντε λεπτά και θα αξιοποιήσω την, ε, το, το σφυράκι μου για να σας διακόψω όταν χρειάζεται. Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας, για την παρουσία σας και τα ξαναλέμε.